Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε Μόνο όμως όταν έρθει να κάτσει εδώ δίπλα, δίπλα μας ο αντιπρόεδρος. Ωραία, ωραία. Σας παρακαλώ καθίστε. Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι αποφάσει των ε, συντονιστών από τι δύο προηγούμενε συνεδριάσει των συντονιστών έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι τι 5 μέχρι τι 3 σήμερα το απόγευμα θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν. Επίση, να σα ότι στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών μιλήσαμε για την εργασία που μπορούν να μας κάνουν οι ε, ομάδες μελέτης, τα τμήματα μελέτης ε, και θέλουμε τις προτάσεις ε, των πολιτικών ομάδων για μελέτες και ενημερώσεις. Μέχρι αύριο είναι η προθεσμία. Παρακαλώ λοιπόν μέχρι αύριο Δεκάτου να στείλετε τις προτάσεις στη Γραμματεία για το τι μπορεί να μας ετοιμάσουν τα τμήματα πολιτικής. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξη και να δώσω το λόγο στον κύριο Βόρθαν από το Ινστιτούτο Fraunhofer για συστήματα ε, καινοτομία Θέλω να τον καλωσορίσω που θα μα ε, μιλήσει για την ενημερωμένη έκθεση για τα, τις για τα μεγάλα προγράμματα TEN-T. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε πρόσωπο. Α, δεν είστε από το Ινστιτούτο Fraunhofer. Α, με συγχωρείτε από το ίδιο λοιπόν τούτο αλλά από άλλο τούτο. Αυτή η ενημέρωση ζητήθηκε από τον προηγούμενο Απρίλιο η προσωρινή εκδοχή της έκθεσης σας αισθάνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Έχετε τυπωμένα ε, αντίτυπα εδώ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να κάνετε Ευχαριστώ κύριε Πράγμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. μαζί με το ΚΙΤ και το PROGNOS, Προκ και εγώ έχουμε από το Ινστιτούτο Φρανχόφερ έχουμε προετοιμάσει από κοινού την έκθεση. Είναι και οι εκπρόσωποι των άλλων δύο εδώ, οπότε μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ποια είναι η δομή της παρουσίασης, ε, τη βλέπετε στη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα θα σας παρουσιάσω τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τις μελέτες περιπτώσεων. Έπειτα θα σας κάνω λόγο για τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, την εκτίμηση του σχεδιασμού και τις μελέτες μεγάλων ε, έργων, κάτι που γίνεται με την ανάπτυξη των υποδομών. Έπειτα θα σας μιλήσω για το σχέδιο, ε, για το πολιτικό πλαίσιο. Και θα ολοκληρώσω με το εκτό σημείο. Ξεκινώ όμω αρχικά με μια ιστορική αναδρομή. Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε την ανάπτυξη αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων. Ήταν μια πολιτική ιδέα, πλέον πρόκειται για μια αναλυτική προσέγγιση. Και έχουμε προτάσει από κάτω προ τα πάνω, αρχικά βέβαια, από τα κράτη-μέλη. τελευταια ομω όμως 5-6 χρόνια και η δική σας Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτά τα δίκτυα για την Ευρώπη και να έχουμε ένα συνολικό δίκτυο διευρωπαϊκών μεταφορών. Επομένως σήμερα έχουμε μια προσέγγιση δικτύου, ολιστική προσέγγιση. Εννέα είναι οι διάδρομοι, όσο το ξέρετε, αυτό τους βλέπετε και στο χάρτη, στη διαφάνεια αυτή. Μ, δεν πολύ καταλαβαίνουμε έτσι, εδώ ίσως είναι πιο απλό. Αυτό λοιπόν το βασικό δίκτυο, όπως είπα, να απαρτίζεται από εννέα βασικούς διαδρόμους. Επιλέξαμε 12 μελέτες περιπτώσεων για την ανάλυση στο πλαίσιο της μελέτης μας, σχεδιασμός, μελέτη κτλ. Πέντε εξ αυτών ε, ήταν πείμα της προηγούμενης μελέτης και έχουμε και νέες πέντε μελέτες περιπτώσεων τις οποίε επιλέξαμε για την προσέγγιση, για την επικαιροποίηση αυτή, αέρον ε, ρήνος, ε, η γραμμή ταχύτητα του Γκάρδι Ούλμ, Λιόν του Ρήνο ε, Γκοτάρδο, Άγιος Γκοτάρδος και ένα τρίτο τούνελ. Αυτά τα περιλαμβάνει αυτή η επικαιροποιημένη εκδοχή. Για κάποια σύντομα στοιχεία το επενδυτικό κόστος είναι από 141 εκατομμύρια 10 δις για τα σχέδια αυτά. Η αξιολόγηση τώρα. Υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ε, το οικονομικό κόστος και το οικονομικό όφελος αυτών των έργων. Αν δείτε δε τους δείκτες είναι από 1,5 έως 2,6 ο λόγος κόστος ωφέλους ε, για τα έργα αυτά. Και αν δείτε και άλλους δείκτες ε, όπως είναι η επιστροφή των πόρων είναι από 25 έως 50 χρόνια. Ποιες ε, ποια είναι τα βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Καθαράς, ε, καθαρά επεξηγηματικά τι γίνεται, ε, πώς λαμβάνονται αποφάσεις για τη συγχρηματοδότηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα έργα, τα project, οδηγούνται σε δράσεις, ενέργειες. Αν δείτε το Rail Baltica, για παράδειγμα, μπαίνουν παραδείγματος σε μια γραμμή στη Λιθουανία και προτείνεται μια ενέργεια για συγχρηματοδότηση ε, για το ΑΙΝΕΑ, τον εκτελεστικό οργανισμό, τον σχετικό, και γίνεται και μία κατάταξη των προτινόμενων δράσεων ανά προτεραιότητα. Και υπάρχει και βέβαια η γάμα δελτα η οποία θα λάβει την τελική απόφαση. Υπάρχουν τέσσερα κριτήρια αξιολόγηση τα οποία έχουμε εδώ ε, λάβει υπόψη μας, ε, τη σημασία, την οριμότητα, τον αντίκτυπο και την ποιότητα. Για να σας δώσω μια ένδειξη για το τι εννοούμε με το πρώτο κριτήριο, σημασία, relevance, έχουμε κάποιους διαγωνισμούς για παράδειγμα για τη χρηματοδότηση και αν ε, σε αυτό το διαγωνισμό μια δεδομένη ενέργεια λαμβάνεται υπόψη. Αν είναι όριμη, οριμότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, διατίθενται ήδη νομικές συγκρίσεις και ούτω καθεξής. Τρίτο κριτήριο είναι ο αντίκτυπος του έργου στο πλαίσιο των κριτήριων αξιολόγησης. Υπάρχει θετική περιβαλλοντική εκτίμηση, είναι καλή η σχέση κόστους-οφέλους, και βέβαια μελετάτε και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου, αν έχει γίνει σωστά ο σχεδιασμός. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο του αντικτύπου, impact, που πρέπει να μελετηθεί σε κάθε δράση και τέλος το ποιοτικό κριτήριο, δηλαδή η διοικητική δομή, αν, είναι τα, αν έχουν τα σωστά σχέδια, εκπονηθεί κτλ. Και Δύο άλλα θέματα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας. Κάποιες φορές τα αντιμετωπίζουν, κάποιες φορές όχι. Διαχείριση κινδύνων, αν χρειαστεί εκ των υστέρων κάποια δράση, τι κίνδυνοι μπορεί να ενέχονται, προσαρμογές και διαχείριση των αλλαγών. Αν υπάρχουν αλλαγές, πώς τις εντοπίζουμε, ποιο είναι το κόστος και πώς θα επηρεάσει αυτό το συνολικό κόστος. Άρα διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αλλαγών είναι άλλες δύο παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη. Τρίτο σημείο, εδώ στον κατάλογό μας, είναι η αξιολόγηση των πολύ μεγάλης κλίμακας έργων, mega project όπως τα αποκαλούμε. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους έργα, Αυτά βέβαια λαμβάνουν ε, και μεγαλύτερο μερίδιο κοινοτική τη τάξεω του 30-40% στα διασυνοριακά και ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τα μία συνοχή κτλ. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ένα τυποποιημένο ε, σύστημα ανάλυσης κόστους ωφέλου, CBA. Βέβαια χρειάζεται και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μεταφορών του παρόντος δεν υπάρχει ένα τέτοιο μοντέλο, τουλάχιστον δεν είναι αρκετά ποιοτικό. Και όταν μιλάμε για αυτά τα πολύ μεγάλης κλίμακας, έργα που κοστίζουν εκατοντάδες, ε, για να μην πω και δις εκατομμύρια ε, ευρώ, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις ευρύτερους, ε, τα ευρύτερα οικονομικά διακυβεύματα. Και το τέταρτο, πάντα χρήσιμο και αναγκαίο είναι να υπάρχουν ανεξάρτητες μελέτες σκοπιμότητας, όχι μόνο αυτές που παρουσιάζουν οι εργολάβοι δηλαδή. Δεύτερο σημείο σε αυτή τη διαφάνεια. Συγχρηματοδότηση μεγάλων, μεγάλης κλίμακας έργων. Βέβαια, αν το μεγαλύτερο μερίδιο, όπως είπα, 40% είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% από κάποια κράτη-μέλη, το μεγαλύτερο μερίδιο το προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να σταθμίζονται πιο καλά και να έχουν μεγαλύτερο βάρος στα κριτήρια τα ενωσιακά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει λόγο εφόσον φέρει και μεγάλο μέρος του κόστους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι αν εξετάζουμε διάφορα σχέδια σε δρόμων υψηλής ταχύτητας σε διάφορα κράτη-μέλη, το κόστος μπορεί να επιμερίζεται μεταξύ τριών παραπάνω χωρών. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και σωστή παρακολούθηση και σωστός λογιστικός έλεγχος. Με την τυποποίηση λοιπόν και την ανάληψη ευθυνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προκύψει εξοικονόμηση κόστους. Τέταρτο σημείο. Μελέτη, σχεδιασμός και οριμότητα των έργων. Βέβαια η μελέτη, ο σχεδιασμός δεν βλέπουμε τη διαφάνεια βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Όχι εκεί. The details, the fourth, point four. Στο τέσσερα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σχεδιασμός λοιπόν. Εδώ πρέπει να οριστούν οι λεπτομέρειες. Δηλαδή αν πρέπει να σεβαστούμε κάποιες προστατευόμενες από περιβαλλοντικής πλευράς περιοχές, ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες, πλοήγηση κτλ, ναυσιπλοήγηση. Θα πρέπει αυτά να μην προκύπτουν στο τέλος μόνο όταν πλέον πρέπει να υλοποιηθεί το έργο, γιατί τότε θα αυξάνεται και το κόστος. Λοιπόν, αν ένα σχέδιο θεωρείται όριμο εάν έχουν οριστεί πρώτον οι διαδρομές, οι ποιοτικές παράμετροι, ποια είναι η ταχύτητα, 180, 220, ποιες είναι οι λωρίδες κτλ. Η σκοπιμότητα επίσης ε, των δομών ε, και των έργων πολιτικού μηχανικού. Πρέπει να ε, δημιουργηθούν τούνελς, γέφυρες και βέβαια και περιβολική εκτίμηση πρέπει να έχει προηγηθεί για να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν. Και νομικές εγκρίσεις. Αν όλα αυτά λοιπόν έχουμε, μπορούμε και αφού βέβαια υπάρχει και μια σωστή εκτίμηση κόστους να λάβουμε την απόφαση το κόστος μπορεί να αυξηθεί βέβαια λόγω κάποιων ασφαλμένων προγραμματισμών ή αύξηση του πληθωρισμού κτλ. Αλλά αυτό είναι κάτι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, και τώρα το πέμπτο σημείο, η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν αυτά τα μεγάλης κλίμακας ε, έργα, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχουμε ένα νέο μηχανισμό που λέγεται ε, πρότυπα για την ε, εφαρμογή των προγραμμάτων Έχουμε λοιπόν ένα τρισδιάστατο μοντέλο υπολογιστή που μας επιτρέπει να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει, πόσο θα κοστίσει και αν πρέπει να προσαρμοστεί ο προγραμματισμός εκτέλεσης, τότε έχεις μία νέα εκτίμηση του κόστους και ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Αυτό επιτρέπει σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να καταλαβαίνουν και τι επιπτώσεις θα έχει η προσαρμογή του προγράμματος ιδίω από πλευράς κόστους. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός, αυτό το εργαλείο μας βοηθάει πολύ. Α, ωραία. Περάσαμε στην επόμενη διαφάνεια. Το πέμπτο σημείο λοιπόν είναι ότι εκτός από την υποδομή πρέπει να δούμε και το πλαίσιο πολιτικής ε, μεταφορών και συγκοινωνιών. Γιατί αυτό αλληλεπιδρά με τις υποδομές ή θα αλληλεπιδράσει. Συνήθως τα μεγάλης διάστασης προγράμματα τα χωρίζουμε σε φάσεις, εφαρμόζουμε την πρώτη φάση, βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η αγορά στον τομέα των μεταφορών, η ζήτηση κυρίως και αν αυξάνεται όπως προβλέψαμε τότε μετά περνάμε στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Αυτό είναι αυτό που προτείνουμε για το διάδρομο Λιόν Τουρίνο. Έχουμε υλοποιήσει την πρώτη φάση, Βλέπουμε πώς εξελίσσεται η αγορά μεταφορών για να δούμε αν θα χρειαστούν οι επόμενες φάσεις. Αυτό μειώνει κάπως τον κίνδυνο υπερεκτίμησης ε, της αύξησης της ζήτησης για μεταφορές. Και υπάρχει και το θέμα της απελευθέρωσης των αγορών μεταφορών με βάση και την ανάπτυξη νέων υποδομών. Για παράδειγμα αυτός ο διάδρομος Λιόν-Τουρίνο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις. Εάν όμως δεν έχουν απελευθερωθεί οι αγορές μεταφορών και στις δύο άκρες της σύραγγας, δεν θα έχουμε τα αναγκαία ωφέλη από αυτό το κόστος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά αυτή, να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός αυτός. Ένα άλλο παράδειγμα όπου οι δέσμοι πολιτικής μεταφορών και δημιουργίες υποδομών πρέπει να συμβαδίσουν είναι το, η σύραγγα gotthard Gotthard-Landsberg. Αποφασίσαμε να χρηματοδοτηθεί από τους φόρους επί των καυσίμων και από τους φόρους επί των βαρέων οχημάτων. Αυτές ήταν οι δύο πηγές χρηματοδότησης. Ήταν λοιπόν ένα συνεκτικό πακέτο ε, πολιτικής υποδομών και μεταφορών. Είναι λοιπόν σημαντικό να ε, αναπτυχθεί σωστά γύρω από την ανάπτυξη των υποδομών και η πολιτική μεταφορών. Το έκτο και τελευταίο είναι το θέμα της συμμετοχής ε, του κοινού. Είναι αναγκαία. Γιατί αν υπάρχει από την αρχή και διαφανώς συμμετοχή του κοινού, θα βελτιώσει την εφαρμογή του, γιατί ακόμη και οι αντίπαλοι ενό τέτοιου προγράμματο μπορεί να έχουν καλέ ιδέε που μπορούν να βελτιώσουν αν εφαρμοστούν το πρόγραμμα και αν ε, εμπλακούν από την αρχή, αποφεύγουμε καθυστερήσει μέσω δικαστικών αφισβητήσεων και αυτό θα μα ε, εξοικονομήσει και χρόνο και χρήμα και δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι το σημαντικό πλεονέκτημα της συμμετοχής του κοινού. Το άλλο παράδειγμα, τα άλλα παραδείγματα είναι ότι μπορεί να γίνουν για παράδειγμα κάποιες ψηφοφορίες για να προωθηθούν κάποια προγράμματα. Το Gotthard Lesberg και πάλι είναι παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκίνησαν με ένα δημοψήφισμα στην ε, Ελβετία για αυτές τις νέες σιδηροδρομικές σύραγγες και μπορεί μεν από οικονομική άποψη να μην δίνουν μεγάλη, ε, μεγάλο κέρδος, αλλά παρόλα αυτά βοηθάνε. Και επίσης ε, η υψηλή ε, δρομική συνδεδρομική σύνδεση Στουτγάρδη-Ούλμα υπήρξαν διαδηλώσεις, καθυστερήσεις που μπλοκάρισαν την ανάπτυξη του προγράμματος και η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία διαιτησίας, συζήτησης με το κοινό για τα υπέρ και κατά και από ό,τι είδαμε υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού, καλή ενημέρωση και στο τέλος η κυβέρνηση ζήτησε να γίνει μια ψηφοφορία που ενέκρινε το πρόγραμμα. Και τώρα μπορεί και πάλι να απεμπλακεί και να προχωρήσει. Οπότε για τόσο μεγάλης κλίμακας ε, έργα πρέπει να γίνονται ή τουλάχιστον συστήνουμε να γίνονται τέτοιες ψηφοφορίες για να υπάρχει διαφάνεια και να προχωρούν τα προγράμματα. Και τέλος, τέλος ε, να αναφέρω μια σύσταση από το πρόγραμμα Netlips, το οποίο πλήρως ε, στηρίζουμε. Εάν ένα πρόγραμμα δεν είναι έτοιμο ή δεν είναι έτοιμο να περάσει στην επόμενη φάση, να το διορθώσετε πριν δαπανίσετε πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντε για την παρουσίαση αυτή. Τώρα έχουμε πρώτα απ' όλα τους συντονιστές αλλά λόγου χρόνου και επειδή έχω ζητήσει πολύ το λόγο, δύο λεπτά παρακαλώ. Βιμ Φαντεκάμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάντε για την αξιοσημείωτη αυτή η παρουσίαση, για τις ε, πληροφορίες, τις αφέστατες, τις οποίες μας έδωσε. Λοιπόν, θα συνεχίσω να μιλάω μέχρι να βρείτε το σωστό κανάλι για τα ακουστικά σας, να ακούτε τη διερμηνία από τα Ολλανδικά. Μία ερώτηση ενδιαφέρεστε εξίσου ε, για τα τοπικά δίκτυα τα οποία θα συνδεθούν ε, με το βασικό σχήμα δίκτυο. Ε, αναφερόμαστε σε διάφορα τοπικά προβλήματα που υπάρχουν για τις διασυνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο. Μας λένε ότι θα υπάρξουν προβλήματα και υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα μεταφορικά συστήματα Έχουμε το σημείο αναχώρησης στο σημείο άφηξης και φαίνεται υπάρχουν κάποια προβλήματα διασύνδεσης. Δεύτερη ερώτηση που αφορά τους πολίτες, τις ανησυχίες των πολιτών. Στην παρουσίαση σας άλλωστε νομίζω ότι αναφερθήκατε σε κάποιες συστάσεις. Έχω την εντύπωση ότι οι συστάσεις αυτές είναι κάπως αδύναμες, πολύ αδύναμες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά χωριά, τοπικές κοινότητες, δήμοι που δεν θέλουν να γίνονται μεγάλα έργα υποδομών. Κοινότητες που ανησυχούν. Ε, τι θα κάνετε για αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν προβλήματα. Ε, ποιες λύσεις μπορούμε να βρούμε. Ανησυχούν περισσότερο οι πολίτες από, από αυτά που μας δώσατε να καταλάβουμε εμείς από αυτά που είπατε. Λάβαμε αυτό το μικρό βιβλιαράκι ε, με τις πληροφορίες και γίνεται διάκριση εκεί μεταξύ των μελετών περιβαλλοντικού αντικτύπου, της, αναλυτικής, ε, της στατικής ανάλυσης αφορά το περιβάλλον, σε επιπτώσει το περιβάλλον και τις μελέτες αντικτύπου για το κλίμα. Ε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η μικροδιάκριση που γίνεται, είναι θεωρητική αυτή η διάκριση, η διαφοροποίηση που γίνεται ή όχι. Και ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες όλων αυτών, αυτό θέλω να ξέρω. Ευχαριστώ Ισμαήλ Χερτοκ. Ευχαριστώ και εγώ τον δόκτορα Σάντε για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δόκτωρα Σάντε, πολλές ερωτήσεις έχω που δεν αφορούν εσάς αμέσως, αλλά τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω όμως ότι είναι παρόντες οι αρμόδιοι από την Επιτροπή. Οπότε θα τις κάνω. Είπατε σωστά, δόκτωρα Σάντε, ότι η συμμετοχή όπως για τη Στουτγάρδη 21, ότι η συμμετοχή των, της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντική. Νομίζω ότι είναι καλό να το ακούσει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον ρωτάω λοιπόν, τα Υπουργεία και δυστυχώς ε, το Υπουργείο Μεταφορών της ε, Γερμανίας φοβάμαι ότι αυτά που αποφασίζουμε εμείς εδώ για τα προγράμματα TENTI δεν τους ενδιαφέρουν και πολύ. Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι πρέπει να εμπλέκονται οι περιφερειακές αρχές. Στη Γερμανία πώς εφαρμόζεται αυτό. Μόνο οι δήμαρχοι συμμετέχουν, ακόμη και αν ε, συμμετέχουν και αυτοί. Δεν συμμετέχουν ούτε καν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, για να μην μιλήσω για συνδικάτα κλπ. Οπότε, ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πίεση μπορείτε να ασκήσετε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για παράβαση, πρώτη ερώτηση, και δεύτερον, τι πρέπει να συμβεί, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ξεκινάει τέτοια διαδικασία παράβασης, τι μέσα έχει να την προωθήσει. Και ξέρετε ότι στην χώρα μου, στην πατρίδα μου, τη Βαβαρία, συζητάμε πολύ για το πότε θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Δηλαδή, είναι δυνατόν να στραφεί η ε, κυβέρνηση κατά της προκήρυξης που έχει γίνει από άλλο φορέα μπορεί να πει όχι δεν με ενδιαφέρει αυτό το πρόγραμμα και είναι δυνατόν εάν αφισβητηθεί να επιστραφούν οι χρηματοδοτήσεις ε, στον κοινό κορβανά Πώς θα καταλάβουμε αυτή την αρχή use it or lose it. Χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα τώρα ή μετά από έξι χρόνια με βάση μόνο τη δική μας απόφαση. Θα ήθελα να μάθω αν έτσι έχει η κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και είμαι και πρώην εισηγητής. Πρόεδρος, εκτός από τους εισηγητές έχω στον κατάλογο Κόλνης, Φαντάλεν, Μπιλμπάο, Μιουρελιέ, Νίλσεν, Εβό, Λιβεράτσκι, Τσούλκα, Αΐντο και Έμπαρ και μετά τον κύριο Ουνίδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κλείσω λοιπόν το κατάλογο τώρα. Ποιο άλλο. Ωραία, κλείνω το κατάλογο. Α, και εκεί. Και εδώ μπροστά. Μάλιστα, μάλιστα, σας είδα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα η Γκεζίνε Μάσνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον δόκτορα Σάντε για αυτή την παρουσίαση. Δεν είναι παρόντες κάποιοι συντονιστές, γι' αυτό έδωσα το λόγο σε εσά κυρία Μάισνα. Ωραία, ωραία, καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Πολλά θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε, αλλά προκαταρκτικά ε, θέλω να μιλήσω για αυτό που είπατε για τη, συμμε... τη σημασία της συμμετοχής της κοινή γνώμης. Βεβαίως, ακριβώς στη Γερμανία, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή, ορισμένα προγράμματα απέτυχαν γιατί δεν συμμετείχε από την αρχή το κοινό. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε, ρωτάω. Πρέπει να συμμετέχει το κοινό σε κάθε πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορούμε για λόγους συμμετοχής του κοινού να αλλάξουμε την σειρά εφαρμογής των προγραμμάτων. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε κανένα πρόγραμμα, αλλά κλασικό παράδειγμα από τη Γερμανία είναι η διαδρομή Y που είναι μέσα στο 10 t Δέκα χρόνια προγραμματίστηκε, δαπανήθηκαν πολλά, δεν συμμετείχαν από την αρχή οι πολίτες, όταν άρχισαν να συμμετέχουν μπλόκαραν το πρόγραμμα. Και ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να διευκολύνουμε την μεταφορά εμπορευμάτων και φοβάμαι ότι αν δεν συμμετέχει σωστά το κοινό μπορεί να προκύψει μπλοκάρισμα. Όλοι λέμε ότι θέλουμε όλο και περισσότερο η μεταφορά αγαθών να περάσει στους σιδηροδρόμους και γι' αυτό προτάθηκε αυτή η διαδρομή Y ε. και τώρα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και δεν βρίσκουμε. Και μέχρι να βρούμε μια σωστή εναλλακτική θα χάσουμε πολλά χρόνια ακόμη και συνεχίζει η μεταφορά εμπορευμάτων οδικός που ούτε αυτό το θέλουν οι πολίτες. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε έγκαιρα τη συμμετοχή του κοινού, πώς μπορούμε να τους ενημερώσουμε για να μην υπάρξει μετά μπλοκάρισμα όταν αντιληφθούν τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Η Μέια Κίλενεν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική των μεταφορών χρειάζεται μακροπρόθεσμο όραμα. Το πακέτο εδώ και χρόνια έχει κολλήσει για τους σιδηροδρόμους και όταν επιτέλους ενεκρίθη όλοι θέλουν να γίνει μια αναθεώρησή του. Όλοι θέλουν να αναθεωρηθεί η δέσμη των μέτρων αυτό το πακέτο. Γι' αυτό θέτω μία ερώτηση που αφορά κυρίως τη Φιλανδία. Θα καταλήξουμε να κάνουμε κάτι ή θα επικεντρωθούμε επί των διαμαχών που έχουμε μεταξύ μας, αντί να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Διότι χρειαζόμαστε αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί συγκεκριμένων τομέων. Εκεί όπου βρίσκονται, αντιμετωπίζονται δυσκολίες. Εκεί που είναι δύσκολη η πρόσβαση. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν από μακρές περιοχές Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά πάνω απ' όλα ε, πρέπει να επικρατεί ειρήνη, ηρεμία στο συνδρομικό δίκτυο. Πήραμε απόφαση όλοι μαζί και θα πρέπει τελικά να στηρίσουμε. Ευχαριστώ Κάι Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Η Γαλλία και η Ιταλία ζητούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως το υπογραμμίσατε κι εσείς, για τη γραμμή Λιόν-Τωρίνο, τεράστιο, γιγάντιο έργο, που ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά τον αντίκτυπο για το περιβάλλον και κυρίως για την δημόσια υγεία. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω ότι ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο της Γαλλίας εξέδωσε στις 20 Οκτωβρίου έκθεση και εκεί αναφέρει και παραθέτω ότι ε, στην πράξη δεν παραμένει καμία πόλη ευρωπαϊκή που είναι αρκετά σημαντική πλευρά πληθυσμού και αρκετά κοντά που να δικαιολογεί μια διασύνδεση λιών ε, το Και θα έχει πολύ μικρό κέρδο κοινωνικο-οικονομικό για τις περιοχές αυτές. Και το ελεκτικό συνέδριο αυτό το επέκρινε στην, ε, το 2012 στην πρώτη απόφασή του. Μικρό το κέρδος το κοινωνικό και το οικονομικό για τη γραμμή Λιών και το χρειάζονται επενδύσει από πλευράς Γαλλίας και Ιταλίας ενώ έχουν δημόσιο έλλειμμα μεγάλο. Και διαρωτώμεθα, λοιπόν για το όλο θέμα. Οι δύο χώρες δεν χρησιμοποιούν τις ε, ανανεωμένες υδρομικές γραμμές, 15 με 20% χρήση έχουμε μόνο. Λοιπόν, και οι στόχοι της Λευκής Βίβλου, οι ευρωπαϊκοί στόχοι της Λευκής Βίβλου θα έπρεπε να υλοποιηθούν αμέσως όσον αφορά τα τοπικά, τις τοπικές διασυνδέσεις. Βασικό ερώτημα, οικονομικά. Συνέχεια αυξάνεται ο προπολογισμό για το έργο αυτό. Έχουμε προβλέψει που έχουν διπλασιαστεί εν σχέση με τι αρχικέ προβλέψει. Μιλάμε για κολοσιαία ε, ποσά, 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να φροντίσει ένα μέρο του μηχανισμού διασυνδέσεων ε, να τεθεί στη διάθεση των υποδομών. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα και ποιες είναι οι λεπτομέρειες οι οικονομικές όσον αφορά αυτό το σχέδιο, αυτό το έργο. Ο κύριος Λούντγκρεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ αρκετά όταν μιλάμε για αυτά, αυτούς τους μεγάλους διαδρόμους και πώς συνδέονται με τα τοπικά δίκτυα. Ε, νομίζω ότι στο τέλος η, ο απλός άνθρωπος τελικά βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Απομονώνεται ο άνθρωπος της υπαίθρου. Εδώ μιλάμε για τιτάνια, πολύ μεγάλα έργα. Τα περισσότερα από αυτά ζητούν τεράστιες δαπάνες που τις πληρώνει ο φορολογούμενος. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά τα χρήματα δεν σπαταλώνται, δεν πηγαίνουν στράφη αυτά που διατίθενται για τα τεράστια έργα. Ε, βέβαια όλοι οι πολίτες ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες οι οποίες ε, συνεχώς αυξάνονται. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρο των συντονιστών. Πολλοί άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα λεπτό θα έχει ο καθένα για να ακούσουμε και τι απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημά μου σε σχέση με τις 12 μελέτες περιπτώσεις που μας παρουσιάσατε από τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των μεταφορών νομίζω ότι μας προκαλούν πιο πολλά ερωτήματα για τη γραμμή Μπέτουβε. Μιλάτε και για μια επόμενη μελέτη. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Είναι κάτι έτοιμο, θα το έχουμε αυτό το έγγραφο στη διάθεσή μας σύντομα και να σας πω και κάτι άλλο. Ότι πήρα το τρένο πέρυσι στην πετούβε γραμμή αυτή συγκεκριμένα, αλλά δεν είχαν μπει οι ράγε στην γαλλική πλευρά. Δεν ξέρω γιατί ακριβώ μιλάτε εσεί. Και κάπου αναφέρεται μία τιμή 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ω κόστο. Θα υπάρξει υπέρβαση αυτού του κόστου. δεν έχω καταλάβει. Αν ναι, πόσο. Μπρόβκα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κατάγομαι από την Κροατία. Άκουσα να αναφέρεται 12 μελέτες περιπτώσεων. Όμως, δεν βλέπω το διάδρομο Αδριατικής Ιωνίου που βρίσκεται στο χάρτη των διευρωπαϊκών δικτύων. Μετά την Τεργέστη πάει από την Κροατία, φτάνει στο λιμάνι του Πλότσε και μετά συνεχίζει, διασχίζει η Κροατία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και φτάνει στην Πάτρα, στην Ελλάδα. Στις 28 ε, Αυγούστου έγινε μια συνάντηση στο Βερολίνο από την αιγίδα της κυρίας Μέρκελ και συμφωνήθηκε αυτή η διαδρομή. Έχω τεχνικής φύσεως ερώτηση. Ποιος αποφασίζει τις διαδρομές, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει επιφορτιστεί με το χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με την εθνική στρατηγική. Ποιος αποφασίζει τελικά για τη διαδρομή, και ποια θα είναι η μοίρα του διαδρόμου αυτού Αδριατικής Ιωνίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επόμενος ο Γιάννης Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από τη Βόρεια Σουηδία. Και ο καθένας βέβαια εστιάζεται στους τοπικούς διαδρόμους. Είναι καλό που έχουμε αυτή την έκθεση. Είναι μια περίοδος που έχουμε μεγάλα προγράμματα, προβλέπονται επενδύσεις μέχρι το 2020, πρέπει να βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα, ποιες συστάσεις θα πρέπει να γίνουν, ποια συμπεράσματα μπορούμε να συναγάγουμε. Νομίζω ότι η έκθεσή σας είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολύ καλή ανάλυση. Μια ερώτηση αφορά την συγχρηματοδότηση. Όσον αφορά το θέμα αυτό, στην πρώτη φάση, στην αρχή ενός προγράμματος, ενός έργου, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να τονώνει, να ενισχύει τη συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι πιο σημαντικό στην αρχή από ό,τι στο τέλος. Και έχω ρώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπορούσαμε να φροντίσουμε ούτω ώστε η χρηματοδότηση να είναι πιο εμπροστοβαρή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις που μας, έδωσαν, ε, που μας έδωσε ο κύριος Άντε. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μελέτη ασχολείται με 12 περιπτώσεις που θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν ως ε, παραδείγματα. Δεν μας είπαν όμως ε, τι κριτήρια λαμβα... μας υπόθηκε, τι λαμβάνουν υπόψη, οι επιπτώσεις, η οριμότητα κτλ. Αλλά μου έλειψε ένα γενικότερο κριτήριο η συνεκτικότητα μεταξύ όλων αυτών των ε, ε, στοιχείων. Έχουμε εγκρίνει τέτοια προγράμματα εδώ και 20 χρόνια. Από το 1994 ξεκινήσαμε. Πριν από δύο χρόνια κάναμε αναθεώρηση και ε, είπαμε ποια από τα προγράμματα αυτά εξακολουθούν να είναι προτεραιότητες διότι δεν έχουν υλοποιηθεί. Είπατε ποια είναι τα πλονεκτήματα της σωστής υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων. Χθες αναλύσαμε μέσω κάποιων μελετών το κόστος της μη Ευρώπης. Και για μένα η ερώτηση είναι τι κάνουμε για να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη να έχουν μια λογική και συνεκτική αντιμετώπιση όταν υποβάλλουν προγράμματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ε, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε στα σύνορά μας, που δεν έχουμε επιλύσει εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα στα ε, σύνορα και έχουμε κόστος 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ λόγω αυτών των προβλημάτων στα σύνορα. Είπατε ότι η Ένωση και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τι ακριβώς εννοείται συγκεκριμένα και τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν κάνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αγγέλα Ίντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε άκουσα την, ε, την λέξη λαϊκή βούληση, ε, δημοφιλία μάλλον τη λέξη. Πώς εκδηλώνεται η αντίθετη βούληση ενός πληθυσμού. Πώς μπορούν αυτοί οι πολίτες να υπερασπίσουν τον εαυτό τους από την εφαρμογή την υλοποίηση του έργου. Αναφέρομαι στη γραμμή Τωρίνο Λιών. Δεν είναι αντίθετοι οι πολίτες μόνο και λόγω διότι είναι, θέλουν να παραμείνει η καθιστική ατάξη αλλά διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για το περιβάλλον. Ε, βρέθηκε αμίαντος και ουράνιο στο όρος ε, σε μεγάλες ποσότητες. Σε περίπτωση λοιπόν όπου υπάρξουν μεγάλα προβλήματα για το περιβάλλον, ε, ποιες δράσεις έχουν προβλεφθεί, μπορούν να προβλεφθούν, να εθετηθούν για να αποφευθεί περιβαλλοντική καταστροφή και στην περίπτωση όπου δεν μπορεί να βρεθεί με συγκεκριμένη λύση μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Ρενό Μιζελιέ. Α, συγγνώμη. Α, ο Μπρούνο Γκόλνης καλύτερα. Μπρούνο Γκόλνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου έρχεται να προσθεθεί στα ερωτήματα της συναδέλφου Καρίμα Αντελή και απευθύνεται κυρίως ε, στη γραμμή Λιών Τωρίνο. Πράγματι είναι ένα ελπιδοφόρο έργο και παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Γάλλου ε, ακούστηκαν πολλά θετικά, υπάρχουν όμως και ανησυχίες. Στο έγγραφο μας παρουσιάζεται ένα ποσοστό αποδοτικότητας 4,72, 5,09. Αυτό, αυτή είναι η ψαλίδα. Εντυπωσιακό, αλλά πού βασίζεστε για αυτή την πρόβλεψη. Δεύτερο και τελευταίο ερώτημα. Αναφέρατε το ενδεχόμενο αυτό το έργο να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Κατάλαβα καλά. Στο τέλος του πρώτου σταδίου θα εξετάσουμε την αποδοτικότητα του έργου και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Δεν καταλαβαίνω. Αν ας πούμε διανοίξουμε τη σύραγγα και δεν μπορούμε μετά να εξασφαλίσουμε τις συνδέσεις, πρόκειται για αστρονομικό έργο που όμως δεν θα έχει μέλλον τελικά. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η βιωσιμότητα και η σκοπιμότητα. Ευχαριστώ και τώρα, Γονόμη Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Δεν θα επανέλθω σε ό,τι είπαν οι συνάδελφοι και για τον κόσμο κτλ. Ε, για το Λιοντορίνο και πολλοί άλλοι μίλησαν, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ. Δεν είναι ένα γαλλοϊταλικό ή γαλλικό πρόβλημα, απλά είναι ένα πολύ σημαντικό σκόμβος για την κυκλοφορία. Ε, θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση και για ε, την ε, ε, μικρότερη επιβάρυνση των οδικών αρτηριών και όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Άκουσα και εγώ πόσο μεγάλος είναι ο προπολογισμό. Αυτό το υπολογισμό κόστους ωφέλους ε, είναι σημαντικό να τον έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Είναι πράγματι τόσο καλή αυτή η αναλογία κόστους ωφέλους, επειδή είναι και μεγάλη επένδυση. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε αυτό. Και επειδή ο πρόεδρος της ε, περιφέρειας Ρον Άλπα, Ροδανού Άλπεων ε, έχει έρθει σε επαφή με τον Ιταλό ομόλογο και θα προσφύγουν στην Ιταλική και στη Γαλλική κυβέρνηση, θέλουν να υπάρξει μια επανεπιβεβαίωση της δέσμευσης. Υπάρχει εμπόδια. Ποιο είναι το βασικό που θα μπορούσε να μπλοκάρει αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Επόμενη, Κριστίν Ρεβού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη αυτή που δίνει σημαντικότατες, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Έχω μια ερώτηση που ξεπερνά το πλαίσιο της μελέτης σας, αλλά πολύ συχνά τίθεται. Το θέμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται και κυρίως συγχρηματοδοτήσεις, συγχρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται από τα κράτη. Στο βαθμό που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης και δημοσιονομικών περιορισμών δεν θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο η μείωση χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων διευρωπαϊκών δικτύων των μεταφορών να λαμβάνουν υπόψη τα, τις, τα ελλείμματα των κρατών μελών. Ε, δεν το έχετε θίξει αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα θέσουμε όλοι μαζί. Ε, ε, ευχαριστώ κύριο Λιμπεράτης και ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. θα ήθελα να μιλήσω για το σημείο 82, 3, 4 και την πρώτη φράση ε, των σχολείων στο κείμενο. Τα κριτήρια για την οριμότητα των προγραμμάτων όσον αφορά το υψηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης. Αν τα κριτήρια είναι πολύ χαμηλά, δημιουργείται ένας κίνδυνος. Αυτό αναφέρει η μελέτη. Αυτό έχει συμβεί ήδη, αν ναι ή όχι, σε ποιο βαθμό. Τα κριτήρια θεωρείται ότι είναι πολύ χαλαρά. Αυτό ε, συνεπάγεται ενδεχομένως αύξηση του κόστους. Και ποιος είναι ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει όσον αφορά τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σάντε, σας ευχαριστώ για την έκθεση που φτάνει την κατάλληλη στιγμή μάλιστα. Έχουμε ξεκινήσει νέες ερωτήσεις και συζητήσεις για τα διευρωπαϊκά δικτύα. 300 δισεκατομμύρια ε, επενδύσεων προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα δίκτυα. Βάσει της εκθέσεως μπορείτε να αξιολογήσετε την ποιότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα σχετικά έργα. Μπορούμε πραγματικά να χρηματοδοτούμε έργα που είχαν κάποια σημασία για την ανάπτυξη όλης της υπήρου μας και για την ανταγωνιστικότητά της. Ή ήρθε η στιγμή να επικαιροποιηθούν τα κριτήρια τους ώστε να είναι σίγουρο ότι τα έργα θα είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή, για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Ντεμόντε. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να στραφώ στην γραμμή Τωρίνο Λιών και να πω ότι ήδη έχουν αντιμετωπιστεί κάποιες διαδικασίες έχουν ε, συζητηθεί θέματα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και υπάρχουν όλα τα χέγγια όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία. Θεωρώ δε ότι αυτή η μελέτη ε, ίσως ε, δημιουργεί, αναφέρεται και σε διάφορα συστηματικά και ευαίσθητα θέματα όπως είναι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες. Δεν ε, εξαντλούνται όμως τα θέματα. Λοιπόν, είναι και άλλο θέμα της διασύνδεσης με τα Βαλκάνια. Χρειάζεται επέκταση των διαδρόμων για να είναι πλήρης η διαδρομή. Τι σκέφτεστε λοιπόν όσον αφορά αυτούς τους διαδρόμους. Θεωρείτε ότι πράγματι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα περνάμε στη γραμμή Y. Εάν καταργήσουμε αυτό το σημείο συμφόρησης, σε τι θα βοηθήσει. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την συμφόρηση στα σημεία ε, Ανόβερο, Αμβούργο και Βρέμι. Επίσης, εφόσον για 20 χρόνια θα, ε, θα φτιάξουμε μία σύραγγα ε, μέσα από τις Άλπεις θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επαρκή και απασχόληση. Και αν θέλουμε κατόπιν να διορθώσουμε και την υπάρχουσα σύραγγα, πόσε θέσει εργασία. Στην Ιταλία έχουμε τρία μεγάλα προγράμματα. Λιόν Τουρίνο, Μπρένερο και Ρότερνταμ Γένουα. Αυτό το αποφασίσαμε το 1996 και δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό. Θεωρείτε ότι μέχρι το 2030 θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα τρία προγράμματα ή πρέπει να καλέσουμε την Ιταλία να θέσει προτεραιότητε ούτω ώστε να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα τρία και όχι και τα δύο και τα τρία να είναι στο, στη φάση του 30-40%. Λοιπόν, για το Λιόν Τωρίνο ποιο είναι το κόστο. Τα 12 δι ή τα 26 που προβλέπονται τώρα. Και μπορεί να περάσουμε και στα 30 40 δι, γιατί είμαι από το Βερολίνο και ξέρω πώ ανεβαίνει το κόστο. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα. Εάν δεν ε, είναι κερδοφόρο πλέον ένα πρόγραμμα, εάν αυξάνονται συνέχεια. Και επίσης το Βερολίνο Μπρεσλάου. Αυτή η διαδρομή με 100 εκατομμύρια θα μείνουν κατά δύο ώρες ε, τη διαδρομή. Γιατί δεν είναι προτεραιότητα αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί θέλουμε να μειώσουμε κατά 1% την διαδρομή από, το, από, τη, από τη Στουτγκάρδη στο Ούλμ. Έτσι έχουμε προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ωραία. Θα μιλήσω γερμανικά λοιπόν τώρα. Γιατί πολλές ερωτήσεις ε, ήταν γερμανικά. Με, μου υποβάλλατε πολύ δύσκολες ερωτήσεις για μια σειρά θέματα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ σωστή διαδικασία για να καθοριστεί το πρόγραμμα TEN-T, δηλαδή η Ευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα των μεταφορών. Υποβλήθηκε αυτό το πρόγραμμα, υπήρξαν και καθευντήρες γραμμές, οπότε τώρα νομίζω ότι η αντιμετώπιση μας είναι τώρα πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν τεράστια πρόοδος έχει σημειωθεί. Και για το θέμα λοιπόν της λογικής και της συνέπειας και της συνεκτικότητας νομίζω ότι τώρα είναι συνεπής η αντιμετώπιση μας. Πολλές ερωτήσεις ε, αφορούν ε, τη γραμμή Λιόν-Τωρίνο. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Υπάρχει ένα σημείο συμφόρησης ε, μεταξύ Λιόν και Τουρίνου για το συνολικό δίκτυο και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι στοιχείο της συνολικής μας αντιμετώπισης. Επίσης ε, έγιναν πολλές ερωτήσεις για λεπτομέρειες του Λιόν Τωρίνο. Βεβαίως έχουμε μελέτη κόστους κόστους-οφέλους και αναφέρθηκα σε αυτήν. Η μελέτη αυτή έγινε από το παρατηρητήριο που ασχολείται με την αποτίμηση αυτής της σύραγγας και ασχολείται με το συνολικό αυτό διάδρομο Λιόν Τωρίνο, 256 ε, ε, χιλιόμετρα συγγνώμη, και πολλά υπόθηκαν για το κόστος 26 δις αφορά συνολικά το διάδρομο, όχι απλώς τη σύραγγα. Έχουμε τώρα λοιπόν αυτήν την σταδιακή υλοποίηση, τώρα υλοποιούμε την πρώτη φάση, όπου φτιάχνουμε αυτό το κυρίως τούνελ που θα κοστίσει 8 με 9 δις από τα 26 δις συνολικά για το διάδρομο και μετά θα ελέγξουμε όταν θα έχουμε αυτό το βασικό τούνελ, τη βασική σύραγγα, θα δούμε πώς εξελίσσεται ε, η κίνηση, να δούμε εάν χρειαζόμαστε και άλλα τούνελ και άλλες σύραγγες, διότι χρειαζόμαστε, έχουν προγραμματιστεί άλλα 4-5 τούνελ ε, μεγάλου μήκους. Πρώτα όμως ναι, ναι, 26, 26 δις διορθώνει ο πρόεδρος. 26 λοιπόν είναι το συνολικό κόστος. Τώρα, η επιβάρυνση, η ενδεχόμενη του περιβάλλοντος, τέθηκε το θέμα του ουρανίου στα πετρώματα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας και Ελπίζουμε ότι θα μειωθούν κατά πολύ, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε εντελώς. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ισχύει αυτό. Πότε θα έπρεπε να συμμετάσχει, να εμπλακεί το κοινό από το 2006-2007 συμμετέχει, γι' αυτό έχει προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα αυτό μέσω αυτού του παρατηρητηρίου όπου συμμετέχουν ε, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και πρωτοβουλίες πολιτών και οι περιφέρειες από την Ιταλική πλευρά αυτή λοιπόν η συμμετοχή οδήγησε να μπορούμε τώρα να μιλάμε για υλοποίηση. Αλλιώ θα είχε εφαρμοστεί μόνο στη Γαλλία όπου υπήρχαν ήδη σύραγγε. Στην Ιταλία δεν υπήρχαν καθόλου. Λοιπόν, για τα επόμενα σημεία. Αυτά ήθελα να πω για την αναλυτική αυτή, αλλά τώρα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Ναι, να μιλήσω για αυτά που είπατε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα δίκτυα δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των μεγάλων προγραμμάτων και ε, μακρών διαδρόμων. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια προγραμματισμού. Αυτό το είχαμε στο Rail Baltica. Θέλαμε να υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα με επιπτώσεις στην περιφερειακή κίνηση και ε, τα άλλα μέσα μεταφοράς. Πρέπει πραγματικά ε, τα προγράμματα αυτά να εντάσσονται στο συνολικό τους περιβάλλον. Παράδειγμα, υψηλής ταχύτητας ε, σιδηρόδρομος Ούλου Στούτκαρτ, πώς συνδέεται με το Στούτκαρτ 21. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία στην έκθεση. Λάβουμε υπόψη τα περιφερειακά δίκτυα. Δηλαδή θέλουμε μεταφορά από σπίτι σε σπίτι, όχι μόνο μέσω του διαδρόμου. λάβουμε υπόψη το συνολικό πλαίσιο ε, σιδηροδρομικών προγραμμάτων το 2004 και έχουμε και εταιρικέ σχέσεις ούτω ώστε να συνεργαζόμεθα και να εγγυόμεθα ότι θα συνδέονται οι διάδρομοι και με τα περιφερειακά δίκτυα και με τα τοπικά δίκτυα. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη συνολικά το δίκτυο, όχι μόνο το διάδρομο, όχι μόνο τις διαδρομές, τις γραμμές υψηλής ταχύτητας. Τώρα, για το θέμα της συγχρηματοδότησης από την αρχή. Ο Γερμανός Υπουργός ε, Μεταφορών έχει μια κυβερνητική επιτροπή συστήση που ασχολείται με τα λάθη του προγραμματισμού. Επειδή είχαμε πολλά προβλήματα και διαπιστώσαμε ότι υπήρξε καταστροφή για τρία μεγάλα προγράμματα, αυτή η επιτροπή προσπάθησε να λύσει τα προβλήματα, να καταδείξει για ποιους λόγους είχαμε αυτή την καταστροφή. Γιατί αυτά τα προγράμματα μπήκαν σε λάθος τροχιά. Ένα ουσιώδης λόγος είναι ότι η προκαταρκτική φάση των προγραμμάτων είναι πολύ αναλυτική και οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση υποθέσεις που ε, δεν ισχύουν πάντα. Έτσι έγινε για αυτά τα τρία προγράμματα. Οι πολιτικές αποφάσεις λήφθηκαν με βάση πολύ πρόορη, ε, σε, με βάση πολύ πρόορη φάση προγραμματισμού και μετά δεν μπορούσε να αναθεωρηθεί. Η συγχρηματοδότηση λοιπόν από την αρχική φάση είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά τον προγραμματισμό, όχι την υλοποίηση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα, να επενδύσουμε περισσότερα. Αυτό ισχύει για όλε τι χώρε. Να επενδύσουμε περισσότερα στην αρχική φάση προγραμματισμού. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερη. Για πολλά προγράμματα ξυπνάμε μόνο όταν ξεκινά η υλοποίηση. Αυτό ήταν το πρόβλημα και με το Στουτγάρδη 21. Οι εναλλακτικέ εξετάστηκαν πολύ αργά μόνο υπό την πίεση των αντιπάλων. Επόμενο σημείο. Ex post ανάλυση. Βεβαίως, ex post έχουμε κάνει μελέτες ε, κόστους οφέλους για να συλλέξουμε εμπειρία για τα μεγάλα προγράμματα. Για κάθε χώρα που έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα είναι μοναδικό. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί ε, τα επόμενα 20-30 χρόνια τόσο μεγάλο πρόγραμμα σε μια χώρα. Οπότε γίνονται μεγάλα λάθη προγραμματισμού γιατί δεν υπάρχει πείρα με μεγάλα προγράμματα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η πείρα που έχουμε συλλέξει από τα μεγάλα προγράμματα να μπορεί κάπου να συλλεχθεί και να μπορεί να αξιοποιηθεί. Για παράδειγμα να έχουμε μια βάση ενημέρωσης με τα αποτελέσματα των παρελθόντων μεγάλων προγραμμάτων για να δούμε για παράδειγμα πόσο υπήρξε υπέρβαση κόστους, πόσο ρεαλιστικές ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, γιατί στην αρχική φάση, επαναλαμβάνω, γίνονται πολύ αισιόδοξε προβλέψεις και εκεί γίνονται τα μεγάλα λάθη. Σε σχέση με αυτό, πρέπει να αναφέρουμε και το πρόγραμμα ελέγχου, controlling, δηλαδή να κάνουμε κάποιες εξομοιώσεις του πώς θα εξαλειφθεί το πρόγραμμα. Αυτό το πρότεινε η Κομισιόν στο Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας γιατί αυτές οι δυνατότητες δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στο παρελθόν. Δηλαδή ένα πρόγραμμα πρέπει να το παρακολουθούμε από την αρχή, μόλις ξεκινήσει να υπάρχει. Να υπάρχει αυτό το BIM, αυτός ο μηχανισμός για την ενημέρωση, για τον έλεγχο, να έχουμε δηλαδή τρισδιάστατη εξομοίωση, ούτω ώστε κάθε λεπτομέρεια να μπορεί να εξεταστεί. Γι' αυτό είναι πολύ ουσιώδες αυτό, γιατί στη φάση προγραμματισμού να, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις. Γιατί αυτές οι τροποποιήσεις είναι που χαροποιούν τόσο πολύ εκ των υστέρων τις κατασκευαστικές εταιρείες γιατί μπορούν να τις υπερτιμήσουν και να έχουμε υπερβάσεις κόστους. Αν έχουμε τέτοια μέσα από την αρχή εξέτασης και ενημέρωσης πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα ελέγχου. Και τελευταίο, για δεν έχουμε πολύ χρόνο πρόεδρε, είναι αυτή, αυτός ο ηθικός κίνδυνος. Βεβαίως ε, οι οικονομολόγοι πάντα το αναφέρουν αυτό. Όταν κάποιος ο οποίος ε, ε, δεν έχει ευθύνη, τελικά παίρνει σοβαρές αποφάσεις, τότε υπάρχουν προβλήματα. Αυτό αφορά τοπικές αρχές, αφορά τις ε, περιφερειακές αρχές, προτείνονται υπερβολικές χρηματοδοτήσεις. Αυτό ισχύει και για ευρωπαϊκής διάστασης ε, προγράμματα. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά προτείνονται υπερβολικών διαστάσεων προγράμματα. Δεν θα πω τώρα παραδείγματα για να μην υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με κάποιες χώρες αλλά θεωρώ ότι κάθε αίτημα που υποβάλλεται για μεγάλο πρόγραμμα πρέπει να ελέγχεται πολύ αναλυτικά να δούμε αν έχει τις σωστές διαστάσεις αν είναι αναγκαίες αυτές οι διαστάσεις ή για παράδειγμα πόση ταχύτητα δεν χρειάζεται παντού να υπάρχουν ε, σειρμοί υψηλής ταχύτητα θα μπορούσαμε να έχουμε και διαδρόμους όπου έχουμε τρένα 160-180 χιλιόμετρων. Αυτό αρκεί για παράδειγμα για μεταφορά ε, εμπορευμάτων. Δεν χρειάζεται να έχουμε παντού την τελευταία λέξη της τεχνικής. Άλλο. Ένα παράδειγμα να αναφέρω το Βερολίνο Σόνεφελ, το αεροδρόμιο, όπου έχει τριπλασιαστεί το αρχικό κόστος. Ξέραμε από τον προγραμματισμό ότι στο τέλος ο φορολογούμενος θα πλήρωνε τα σπασμένα. Αν ήταν ιδιωτικό το πρόγραμμα, σίγουρα θα είχε ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Γιατί πολλά τα οποία συμπεριλήφθηκαν στον πραγματισμό δεν χρειάζονταν. Ήταν υπερβολικά. Και έγινε τόσο περίπλοκο το πρόγραμμα που κατέληξε να είναι και τόσο ακριβό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ουνίτη να αναφέρω το εξής. Η διαδρομή Βερολίνο-Αμβούργο έχει υψηλότατη ταχύτητα 240 και η κολονία, κολονία Φραγκφούρτη έχει, έχει μέγιστη ταχύτητα 300 χιλιόμετρα. Φυσικά η μέση ταχύτητα είναι 195 από την άλλη μεριά μεταξύ κολονίας και ε, ε, Φραγκφούρτης ενώ η μέση ταχύτητα μεταξύ ε, Αμβούργου και τη άλλη πόλη, Βερολίνου και Αμβούργου, είναι 198. Άρα δεν είναι η μέγιστη ταχύτητα το σημαντικό, αλλά η μέγιστη ταχύτητα και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα τη δυνατότητα να λάβω το λόγο στο πλαίσιο τη συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για μια πολύ ποιοτική μελέτη, οφείλω να το πω αυτό. Ουσιαστικά είναι η συνέχεια μιας μελέτης που είχε διενεργηθεί ήδη το 2013 και θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά την εξαιρετική ποιότητα των συστάσεων που μας παρέχονται. Είναι άκρος αντικειμενική, αμερόληπτη αυτή η μελέτη και προσβλέπουμε βέβαια στη συνέχιση της συνεργασίας μας και με τα συμβουλευτικά γραφεία, τα μελετητικά αυτά γραφεία για να υλοποιηθούν αυτές οι συστάσεις. Νομίζω ότι Στη μελέτη αυτή γίνεται πολύ καλή διάκριση μεταξύ των βελτιώσεων που ήδη είναι ορατές και έχουμε και τον νέο κανονισμό και το ΣΕΦ και βέβαια έχουμε και τους τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτούνται ή τέλος πάντων θα ήταν απαραίτητες περισσότερες βελτιώσεις. Να σχολιάσω κάποιες ε, κάποιες παρεμβάσεις πολύτιμες από τους βουλευτές. Πρώτον, πολλοί βουλευτές επισήμαναν ε, μια δυσκολία που παραμένει ή πώς θα πειθαρχήσουν οι εθνικές αρχές και θα εξασφαλίσουν ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν τελικά είναι ακριβώς αυτά που επιθυμούσαμε. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά γιατί πρώτα απ' όλα μας δώσατε τη δυνατότητα να έχουμε τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά και τον κανονισμό ΣΕΦ, δηλαδή τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Και έχουμε και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και το είδος των έργων που εξετάζουμε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο, για πρώτη φορά ξεκινούμε πλέον πάρα πολύ αναλυτικές και διαμακρών συζητήσεις με εθνικές τοπικές αρχές ουσιαστικά για να προετοιμάσουμε ε, την ε, υποβολή σχεδίων. Συζητούμε με τις διάφορες αρχές και ελπίζουμε ότι αν αποδειχθεί ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, αυτό θα βοηθήσει περισσότερο και πιστεύω ότι θα το ξέρουμε αυτό όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης ε, την δυνατότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, είπα και ο κύριος Σερτούκ. Ξέρετε, δύσκολα μπορούμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη κατά συγκεκριμένων αρχών γιατί δεν πρότειναν ή δεν προώθησαν το σωστό έργο. Αλλά μπορούμε να κατανείμουμε τους πόρους στα σχέδια που θεωρούμε ότι έχουν τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Και αυτήν την έννοια είναι πολύ εύγλωτο το, η μελέτη, τα απορίσματα της μελέτης χρησιμοποιούμε αυτά τα νέα κριτήρια αξιολόγησης. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της ποιότητας του κάθε έργου. Ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρθηκε είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για μια πιο εμπροστοβαρή χρηματοδότηση των έργων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα θυμάστε όταν συζητήσαμε με τον πρώτο διαγωνισμό, συζητήσαμε και μαζί σας το ενδεχόμενο να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 12 δισεκατομμύρια μάλιστα είχαμε θέσει επιτάπητος τότε, δηλαδή το ίμιση του επιτάητους προπολογισμού. Και αυτό το είπαμε γιατί ο στόχος ήταν έστω ε, με αλλά με αποφασιστικό τρόπο να συνεισφέρουμε σε αυτή την εμπροστοβάρη χρηματοδότηση πολλών έργων για να βοηθήσουμε στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης ο διάδρομος Ανδρετικής Ιωνίου. Είναι μια πρωτοβουλία αλλά δεν είναι ακόμη γεγονός υπό την έννοια ότι δεν έχει ενταχθεί ε, στα διευρωπαϊκά ακόμη, όπως είπατε. Τα καλά νέα βέβαια είναι ότι φυσικά και επεξεργαζόμαστε τα του εν λόγω διαδρόμου, γιατί είναι μια πολύ σημαντική επέκταση του υφιστάμενου δικτύου που θέλουμε να αναπτύξουμε. Η πολύ καλή είδηση είναι ότι στο Βελιγράδι πριν από δύο εβδομάδες ανακοινώσαμε επισήμως σε υπουργική συνάντηση ότι θα ξεκινήσουμε τώρα τις εργασίες για την επέκταση του διαδρόμου αυτού προς τα Δυτικά Βαλκάνια και με την ίδια μεθοδολογία αλλά και ε, με τους ίδιους συντονιστές. Άρα είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει συνέχιση και θα έχουμε πολύ ομαλή εξέλιξη για την ένωση αυτών των διαδρόμων. Ο πρόεδρος ε, δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσετε. Μάλιστα. Ε, το επίκεντρο, η εστίαση ε, στα μεγάλης κλίμακας έργα. Πράγματι υπάρχει αυτή η εστίαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι τελικά τα μεγάλα αυτά έργα ούτε ε, το 20% της συνολική χρηματοδότηση από το Connecting Europe δεν θα πάρουν δυνητικά. Είναι περιορισμένο το εύρο. Ε, το υπολογίσετε, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση συνοχής, μιλάμε για 10% χρηματοδότηση που δυνητικά πηγαίνει σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ευχαριστώ. Να πω το εξή το τελευταίο. Ξέρω ότι ο μέσος όρος είναι γύρω στο 10%. Ορισμένε φορές είναι 20%. Αλλά επειδή κοστίζει 26 δισεκατομμύρια το Λιόν Τωρίνο, αποφασίσατε ε, ήδη ένα κόστος και μετά είπατε ε, δεν πειράζει να αυξηθεί γιατί θα τα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Κομισιόν. Είπε τι σημαίνει αυτό. Είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέτε. Δεν πρόκειται να σας ε, δώσουμε τόσο πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Βεβαίως πολλοί επιθυμούν πολλά αλλά δεν επιτυχάνουμε πολλά. Αυτό θέλουμε να δούμε και στη συνέχιση τη συζήτηση. Για τα μεγάλα προγράμματα θα έχουμε βέβαια πολύ χρόνο και γι' αυτό ευχαριστώ πρώτα απ' όλα θερμότατα τον κύριο Σάντα και τον κύριο Ρότενβέρτερ για τη μελέτη. Ακούσατε και πολλούς επένους από άλλους για την μελέτη σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην περαιτέρω εργασία σας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και περαιτέρω τη συζήτηση αν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς το μικρόφωνο του Πρόεδρου είναι κλειστό. Το μικρόφωνο του Πρόεδρου είναι κλειστό. Το μικρόφωνο του Πρόεδρου είναι κλειστό. Αν μπορεί κανείς να του πει να το ανοίξει. Α, με συγχωρείτε, τώρα ο Πρόεδρος. Λοιπόν, υπάρχουν ε, ε πολλές περιπτώσεις όπου ε, καταργούνται πολλά τρένα, ιδίως νυχτερινά τρένα ορισμένες φορές αντικαθιστώνται με ε, λεωφορεία, με πούλμαν και σε άλλες περιπτώσεις δεν αντικαθιστώνται. Αυτό απασχολεί πολύ την ε, Γερμανία, για να εφερθεί στο Κοινοβούλιο. Έχουν υπογραφεί ε, πολλές, πολλά αιτήματα. Όταν καταργήθηκε για παράδειγμα η, γραμμή μεταξύ, η νυχτερινή γραμμή μεταξύ Βερολίνου και Βρυξελών Έξι εβδομάδε πριν την κατάρριξη σταμάτησαν να κλείνουν θέσει χωρί να πούν τίποτα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο σε εκπροσώπου τη Κομισιόν, σε εκπροσώπου των σιδηροδρόμων και εκπροσώπου των επιβατών των σιδηροδρόμων να μιλήσουν για το θέμα αυτό από πέντε λεπτά και μετά θα κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα με τα μέλη. Και ο πρώτο ομιλητή, όπω ήδη ακούσαμε, είναι ο Όλιβερ Ονίδη που είναι διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση MOVE μεταφορών. 10 λεπτά κύριε Ονίδη, έχετε το λόγο γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, δύσκολο. Βέβαια, τελικά η απόφαση να ανοίξει ή να σταματήσει μια υπηρεσία όταν δεν ανήκει σε υποχρέωση του δημόσιου τομέα, η απόφαση βασίζεται σε εμπορικά κριτήρια. Αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετές πτυχές που μπορούμε να επεξεργαστούμε με την υποστήριξή σας, ούτω ώστε στο βαθμό του δυνατού να παρέχουμε αυτού του είδους υπηρεσίες. Πρώτη πτυχή που θέλω να αναφέρω. Η εικόνα τελικά δεν μπορεί να θεωρηθεί λευκή ή μαύρη. Και αυτό το βλέπουμε από την έκθεση την πρόσφατη που δημοσιεύθηκε πριν από έξι μήνες που αφορά την αγορά και τα στοιχεία δείχνουν ότι σε αρκετές διαδρομές, σε αρκετές χώρες η διακίνηση διεθνή των επιβατών έχει αυξηθεί και έχει αυξηθεί και το είδος των υπηρεσιών παρέχεται, αυξηθεί ο αριθμός των ειδών υπηρεσιών. Θα αναφέρω τέσσερις τομείς όπου χρήζουν βελτιώσεων. Πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν είναι αποδεκτό σήμερα να χρησιμοποιούμε στοιχεία που χρονολογούνται από το 2012. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βελτιωθεί μέσω εφαρμοστικής πράξης, κάτι που προβλέπεται στην ε, επανεξέταση του όλου συστήματος που εκεί αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να αποστέλλονται στο Eurostat και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να γίνεται πιο σωστή εκτίμηση της ε, εξέλιξης αγοράς και τη δυναμικότητα αγορά των σιδηροδρόμων. Δεύτερον, πρέπει να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο. Αυτή η συζήτηση είναι στο επίκεντρο του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους, θέμα που ακόμα συζητείται. Ξεκίνησαν συζητήσεις, είναι πολύ αποδοτικές όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών και βέβαια θα πρέπει να ανοιχθεί αγορά και για τους ε, επιβάτες του εσωτερικού και είναι κρίσιμη σημασίας διότι η διεθνής κυκλοφορία δεν μπορεί να ιδωθεί απομονωμένα, πρέπει να θεωρηθείτε αποτελεί τμήμα του ευρυτέρου δικτύου και έτσι χρειάζεται να δώσουν περισσότερες υπηρεσίες τους επιβάτες εσωτερικού και αυτές οι υπηρεσίες θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών για τους επιβάτες υιοθετώντας το μοντέλο του τομέα των αερομεταφορών. Θα πρέπει να επιταχυνθούν τρίτον ε, κάποια εργαλεία που αφορούν τους χρήστες, τους καταναλωτές. Έχουν γίνει καλές προσπάθειες στο TAP TSI, δηλαδή προδιαγραφές που απαιτούνται ούτω ώστε ταχύτερα να χορηγούνται υπηρεσίες, να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα έκδοση εισιτηρίων, αλλά και προγραμματισμός ταξιδίου, ούτω ώστε να μπορούμε να διαφημίζουμε και καλύτερα διάφορες υπηρεσίες και οι χρήστες να μπορούν να πάρουν μια απόφαση πλήρως ενήμερη. Αυτή είναι και συνεχής ε, απέτηση και του Κοινοβουλίου και τους επόμενους μήνες ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό υλοποιήσεως αυτών των μέτρων. Τέλος, έχουμε τις υποδομές. Το συζητήσαμε αυτό προηγουμένως. Με τα νέα εργαλεία, με τα προγράμματα εργασιών που αφορούν τους διαδρόμους και την έμφαση που δίδεται επί τεχνικής διαλειτουργικότητας με τα διάφορα συστήματα όπως το RTMS με όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα προσθέσουμε ένα άλλο θετικό στοιχείο, τόσο ώστε τα, οι διεθνείς μεταφορές σιδηροδρομικές να γίνουν πιο ελκυστικές και να διευκολυνθούν αυτές οι υπηρεσίες από τεχνική σκοπιά και να μειωθεί και το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Λίμπε Λόχμαν από το CER. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να έχω τις διαφάνειές μου στην οθόνη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα, δίνετε δυνατότητα στο CER να εκφράσει και την άποψη της κοινότητας που εκφράζει και τις επιχειρήσεις συνδρομικές και όχι μόνο την πλειοψηφία των επιβατών στα τα, τα γρήγορα τρένα, αλλά και τα νυχτερινά τρένα. Η συνομοσπονδία μας εκπροσωπεί τις περισσότερες εταιρείε τις εταιρείε ε, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εκπροσωπούμε τη φωνή ε, όλου του τομέα εν γέννη. Θα αναφέρω κάποια στοιχεία στην αρχή. Πιστεύουμε ότι σίγουρα οι σιδηρόδρομοι αποτελούν τη λύση για τις μεγάλες προκλήσεις που θα πρέπει να αναμένονται από τη μελλοντική ζήτηση όσον αφορά την κινητικότητα και από την σπάνιδα ε, των πόρων, κυρίως πλευρά των ορυκτών καυσίμων και του πετρελαίου στο μέλλον και επίσης και συμφορήσεις και από την πλευρά των οδικών δικτύων καθώς και των εθέρων, διότι ε, θα έχουμε επίσης προβλήματα και πλευράς αερομεταφορών. Λοιπόν, οι σιδηρόδρομοι που χρησιμοποιήσουν τη λύση και πιστεύουν οι σιδηρόδρομοι πραγματικά μπορούν να παράσχουν τη σωστή απάντηση στις προκλήσεις. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω και κάποια στοιχεία. Λοιπόν, ποιο είναι το ποσοστό διακίνηση εσωτερικού και διεθνεί μεταφορέ όσον αφορά του επιβάτε χιλιόμετρα. 94% είναι στο, τομέα του εσωτερικού, 6% στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, θα αφορούν τι διεθνείς υπηρεσίε αυτό είναι η διαχωρισμό μεταξύ ε, μεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού. Όσον αφορά μακρέ αποστάσει και περιφερειακέ αποστάσει, βλέπετε 50% περίπου είναι περιφερειακέ αποστάσει, 25% περίπου ένα τέταρτο είναι διαδρομέ υψηλή ταχύτητα και άλλο ένα τέταρτο είναι μακρά απόσταση. Τα ποσοστά αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μα όταν αναφέρουμε ε, τι δυνατότητε που παρέχονται διεθνεί μεταφορέ διαδρομικέ. Ποιε είναι οι προκλήσει ε, θα ξεκινήσω με τις ε, τεχνικές προκλήσεις από την έποψη όχι μόνο των ε, τρένων υψηλής ταχύτητας που έχει αυξανόμενο δυναμικό τομέα, αλλά τεχνικές προκλήσεις που αφορούν την αποδοχή και την αδειοδότηση των διαφόρων οχημάτων επεμβατών Λοιπόν, έχει καταληφθεί το καθεστώς RSI και έχει δημιουργηθεί κάποιο κενό που θα πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για μελλοντική απρόσκοπτη κυκλοφορία των διαφόρων βαγονιών των επιβατικών. Όπως αναφέραμε, διεθνείς αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται επιβορικής βάση, οπότε ε, πρέπει να υπάρχει κέρδο για να υπάρχει σωστή ποιότητα των υπηρεσιών και άλλε παράμετροι συζητήθηκαν το πρωί και αναφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τι μικρές υποδομέ, ε, μικρέ επενδύσεις για τις υποδομές των ιδιοδρόμων που επηρεάζουν τους ιδιοδρόμους και δεν υπάρχει ισότιμο ανταγωνισμό, και αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης. Λοιπόν, πρέπει να εστιαστούμε στις νυχτερινέ ε, υπηρεσίες ε, και εσείς το αναφέρατε Πρόεδρε. Βλέπετε ότι καταλείπονται αυτές οι υπηρεσίες. Βέβαια, ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν προσδοκίε πλευρά επιβατών όσον αφορά την ποιότητα των νυχτερινών τρένων, όσον αφορά την ποιότητα των χώρων φόρτωση των τερματικών, την ποιότητα στα τρένα όπω ε, στα εστιατόρια, ε, τα ντου ε, και κυρίω στι διαδρομέ που διαρκούν 6 με 7 ώρε. Όχι τόσο γρήγορα, παρακαλεί ο Πρόεδρο. Εντάξει, εντάξει. Προσπαθώ να μιλήσω μέσα στα χρονικά περιθώρια που δοθήκα, αλλά μπορούν να, να μεταφράζονται λέει και ο, ο πρόεδρος. Λοιπόν, οι συγκεκριμένε προκλήσει για τα νυχτερινά τρένα. Λοιπόν, να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε των επιβατών. Εν πρώτη, υπάρχουν αυξανόμενε πιέσει λόγω τη αύξηση της ε, τη κυκλοφορία των ε, αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστου. Λοιπόν, ο ανταγωνισμό είναι πολύ δύσκολο στι κοινέ υπηρεσίε. Μετά από το πλευρά συνδρομικού δικτύου θα πρέπει να λειτουργούν τα τρένα, κυρίω τα νυχτερινά τρένα, κατά τη τη νύχτα και οι νυχτερινέ ώρε χρησιμοποιούνται περισσότερο για την συντήρηση του δικτύου και για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα πώ να βρούμε ε, τη δυνατότητα διαδρομών. Και μετά είναι και το θέμα του συνδρομικού υλικού. Για τα νυχτερινά τρένα χρειαζόμαστε ειδικά τρένα με κρεβάτι ε, λοιπά Και είναι συγκεκριμένε ανάγκε και δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα βαγόνια την ημέρα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χρήση αυτών των βαγονιών. Μετά υπάρχει ανταγωνισμό με τι ε, αεροπορικέ εταιρείε χαμηλού κόστου και αυτό είναι κάτι που εμποδίζει την εμπορική ελκυστικότητα των επιβατικών υπηρεσιών σε διεθνείς μεταφορές και κυρίως ε, στα νυχτερινά τρένα θα πρέπει να εντοπίσουμε τη σωστή λύση γι' αυτό και η σωστή ε, λύση κατά την άποψή μας είναι οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας όπου εκεί υπάρχει μεγάλο δυναμικό για να αποφύγουμε και τις συμφορήσεις σε νέε μεταφορές και να ε, βελτιωθεί η συνοχή ε, μεταξύ των χωρών και γενικά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Αναφέρθηκε τώρα ισότιμος ανταγωνισμός, οι δίκαιες συνθήκες, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το σημαντικότερο πέρα από τη διθεσιμότητα των διαδρομών ε, και αυτό είναι που μπλοκάρει την εμπορική βιωσιμότητα. Πρέπει να εξορροπήσουμε τις, ε, τις υποδομές, τα τέλη, το ΦΠΑ και εσωτερική ύψη του εξωτερικού κόστου αν θέλουμε να προσθέσουμε στις διεθνείς μεταφορές και τις νυχτερινές μεταφορές, τα νυχτερινά τρένα, ε, δυνατότητα κέρδους. Στο τέλος, αν μιλήσουμε για το μέλλον των σιδεοδρόμων θα πρέπει να καθορίσουμε το προφανές, δηλαδή ότι έχουμε 100% του, ότι καταβάλουν τέλη 100% στο συνδρομικό δίκτυο τα τρένα και 0,9% στις οδικές μεταφορές. Λοιπόν, έχουμε ένα όραμα, τι μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά τη μεταφορά των επιβατών. Θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο διεθνείς υπηρεσίες διεθνών μεταφορών. Θέλουμε να αλλάξουμε την προσφορά που παρέχεται και να προωθήσουμε και τις ε, υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, να θεωρηθεί μια υπηρεσία που είναι φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη και θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών με πολυτροπική μεταφορά. Ε, συνεργασία με μεταφορά μέσω λεωφορείων και με αερομεταφορές και να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Ευρώπης με τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιβατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω ότι χαιρόμαστε πολύ με την ευκαιρία που έχουμε και εμείς να συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Διαφάνεις δεν έχουμε. Εν συντομία θα σας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών εκπροσωπεί 35 οργανώσεις ε, για τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών σε 20 ευρωπαϊκές χώρες η ανάγκη να είναι εύκολες ε, οι συνδρομικές μεταφορές ήταν και ένας λόγος που μας εισπήρωσε και δημιουργήσαμε αυτή την Ομοσπονδία πριν από 20 χρόνια. Πρώτον, το θέμα της επιλογής. Είναι σημαντικό οι επιβάτες να μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο της ε, μεταφοράς τους για τα διεθνή τους ταξίδια. Και θα πρέπει να αναγνωρίζουν οι επιλογές και τα περιβαλλοντικά πλονεκτήματα του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει όμως να είναι δυνατόν να παρέχεται και μια ελκυστική υπηρεσία σε προσιτή τιμή. Αυτό εφαρμόζεται στα διεθνή ημερήσια τρένα, αλλά και στα διεθνή βραδινά, νυχτερινά τρένα. Δεν θέλω να κάνω διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και διεθνών σύρμων. Οποιοδήποτε τρένο συνδέει δύο ή περισσότερες ε, χώρες θεωρείται διεθνές, διεθνής σύρμος. Είναι γεγονό ότι ο ανταγωνισμό μεταξύ σιδηροδρομικών και άλλων μεταφορών δεν είναι θεμητό. και συμφωνούμε με τον δόκτωρα Λόχνερ και του ε, συναδέλφους του από την Συνομοσπονδία ε, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Όμω, οι χαράκτε πολιτική και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι επαγγελματίε του κλάδου σιδηροδρόμου τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν τα πράγματα. Η εμπειρία πολλών οργανώσεων μελών μα δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερο διάλογο και μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ ε, των εθνικών διαχειριστών υποδομών. Θα πρέπει η πρόσβαση ε, στις συνδεδρομικές υπηρεσίες ε, να μελετηθεί. Πρέπει να, είμαστε, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ό,τι αφορά ε, τη, τα τέλη. Ε, θα πρέπει και ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη τη διασυνοριακή και την εθνική κυκλοφορία. Η χρηματοδότηση. Αν ένας διαχειριστής λάβει δημόσια χρηματοδότηση, δεν θα πρέπει ε, να υπάρχει προϋπόθεση διατήρησης διασυνοριακών μεταφορών, αν χρειάζεται, όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη νύχτα, αν αυτό αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σίγουρα και οι δύο πλευρέ μπορούν να κερδίσουν. Οι πολίτε έχουν μεγαλύτερη επιλογή που να ζήσουν, να δουλέψουν, να σπουδάσουν. Είναι πιο εύκολη επίση ε, η μεταφορά από τη μία περιοχή στην άλλη και για λόγους αναψυχής και αυτό βοηθά την τοπική οικονομία. Θα πρέπει βέβαια ε, να πιστούν οι αρχές. Ε, υπάρχει ένα, μια, ένα γύρο τραπέζια, στρογγυλό τραπέζι που κάνει πολύ καλή δουλειά, στηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πρέπει να πω ότι και τα περιφερειακά κονδύλια ήταν πολύ σημαντικά ε, για τη σχέση Βίλαχ-Ούντινε και τη σύνδεση πραγματικού χρόνου. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση και στήριξη περισσότερων τέτοιων έργων για τη διασύνδεση μεταξύ των πόλεων βοηθά ε, και τις ε, μετακινήσεις των πολιτών, τις διασυνοριακές όταν υπάρχει franchising. Το τροχαίο υλικό θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Από την Τσεχική Δημοκρατία μέχρι τη Γερμανία υπάρχει μια γραμμή ε, πολύ καλής ε, συμφωνίας δικαιόχρησης franchise. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και ο τεχνικός πυλώνας του ατρασυνδεραμικού πακέτου. Προσβλέπουμε σε αυτό και κάθε νομοθεσία θα πρέπει να διέπεται από δύο κριτήρια. Αν θα ωφελεί τους επιβάτες και αν θα διευκολύνει τις διεθνείς συνδεδρομικές μετακινήσεις. Ό,τι αφορά τα νυχτερινά τρένα. Για τα διεθνή νυχτερινά τρένα υπάρχουν και, άλλοι, ε, και άλλες παράμετροι. Δηλαδή, εάν είναι λογικές οι ώρες όποιες λειτουργούν, εάν είναι ε, το ταξίδι εύκολο, αν υπάρχει κουκέτα μπορεί να κοιμηθεί δηλαδή ο ταξιδιώτης ε, και αν υπάρχει σχέση και πρόσβαση με τα πρωινά. Είχα φτάσει 7 το πρωί στο Μόναχο με ένα ε, νυχτερινό τρένο, είχα αργήσει και θα έχανα την ανταπόκριση με το ημερίσιο που όμως περίμενε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η ομαλή σύνδεση νυχτερινών με ημερίσια τρένα. Τώρα, θεωρούμε ότι έχουν ρόλο τα διεθνή νυχτερινά τρένα. Βέβαια ο ρόλος τους δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με το ρόλο που είχαν πριν από 30 χρόνια. Εμείς λοιπόν στην Ομοσπονδία μας ε, απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει μια ανεξάρτητη εξεταστική μελέτη που θα διερευνήσει τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουν τα διεθνή ε, νυχτερινά τρένα για τους πολίτες και να συσχετίσει τα ωφέλη με το κόστος. Γιατί αυτό είναι κλειδί για να προσδιορίσουμε και τη μελλοντική εξέλιξη στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θα ήθελε παρακαλώ να πάρει το λόγο, ορισμένοι ήδη τον έχουν ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον δόκτωρα Λόχμαν διότι και, από, και τον ε, εκπρόσωπο των επιβατών ε, πολύ ενδιαφέρουσες προφορίες δύο ερωτήσεις. Αφορά τη σχέση μεταξύ αυτού του σημείου ε, τη ημερήσια διάταξη και του τέρτου πακέτου ε, σιδηροδρομικών μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά την διακυβέρνηση. Επαρκεί αυτό το τέταρτο πακέτο, δηλαδή. Αν συγκρίνουμε την πληροφόρηση που μόλις λάβαμε με αυτά που ξέρουμε για το πακέτο, θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν περαιτέρω αιτήματα. Επίσης, ποια είναι η σχέση μεταξύ των ε, παρεμβάσεων που μόλις ακούσαμε και του κυβερνητικού τμήματος του σιδηροδρομικού πακέτου. Και μία άλλη ερώτηση. Ανταγωνισμός μεταξύ νυκτερινών ε, σιδηροδρόμων και ε, εταιριών, αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Την προηγούμενη Παρασκευή Καταργήθηκε μία ε, νυχτερινή γραμμή μεταξύ Φραγκφούρτη και Άμστερνταμ γιατί δεν υπήρχε επαρκή ζήτηση. Αυτό το περιέγραψε ο κύριο Λόχμαν και είναι όντω πραγματικό αυτό ο κίνδυνο. Έχω την εντύπωση και μάλιστα σε μια ε, εκδήλωση όπου συμμετείχαμε σε ένα γεύμα μας είπε ένας εκπρόσωπος των ε, γερμανικών σειροδρόμων ότι τα νυχτερινά δρομολόγια δεν είναι κερδοφόρα διότι είναι πολύ ψηλό ανταγωνισμό από τι ε, αεροπορικέ εταιρείε χαμηλού κόστου. Όμω εδώ στην παρουσίαση μου είπατε ότι υπάρχει ε, θετική προοπτική. Τι βάση έχετε για την ε, αισιόδοξη αυτή αντιμετώπιση σα, η Λούση Άντερ. Ευχαριστώ να συγχαρώ τον πρόεδρό μα, τον κύριο Κρέμερ, που εξασφάλισε η περίπτωση του σημείου αυτού στην ημερήσια διάταξη. Είναι σημαντικό το θέμα, πάρα πολύ. Ε, διαφωνώ κάπως με τον κύριο Βαντερ Κάμπ για το θέμα της βιωσιμότητας. Αυτό δεν εξετάζεται αρκετά λεπτομερώς και δεν τονίζεται επαρκώς η πολιτική βούληση και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις που νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνομοσπονδίες σας θέλουν να απαντήσουν και θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως ε, το, αυτά που είπα εκπρόσωπος του EPF, δηλαδή αυτά που είπαν εκπρόσωποι δηλαδή που ζητούν να γίνει μια μελέτη ανεξάρτητη για διαπίστωση των πραγματικών στοιχείων. Και θα πρέπει ε, τις να εξετάσει αυτή η Επιτροπή, τις προδιαγραφές για την ανάθεση αυτής της μελέτης. Πέραν αυτού, τα θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα είναι σημαντικά, αλλά δεν συγκρίνουμε παρόμοια πράγματα. Υπάρχει περιβαλλοντική και πολιτική ανάγκη σχετικά με τι επιθυμίε των επιβατών για τη μετώπιση τη αλλαγή του κλίματο, ώστε να διατηρηθούν οι διασυνοριακέ υπηρεσίε και οι νυχτερινέ υπηρεσίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μα πει γιατί ο κανονισμό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και ο κανονισμό για τη σύνδεση τη Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα κριτήρια ώστε οι υπηρεσίε για τα νυχτερινά τρένα να έχουν προτεραιότητα. Σημαντικότατο θέμα η Deutsche Bahn δεν έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αυτά τα τρένα. Έχουμε στοιχεία των υπηρεσιών της Κοπενχάγης που δείχνουν ότι είναι δημοφιλέστατα τα τρένα και δεν υπάρχει λόγος που να μην μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο. Και άλλες νυχτερινές υπηρεσίες στην Ευρώπη δέχονται επενδύσεις. Από Μόναχο πήγα στο Ζάγκρεμπ έχει νέα τρένα αυτή η διαδρομή και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα υπηρεσιών που λειτουργούν και επιθυμούν να έχουν τι υπηρεσίε αυτέ οι επιβάτε. Άρα δεν πρέπει να εξετάζουμε το θέμα μόνο από εμπορική ε, πτυχή, ε, εμπορική σκοπιά, αλλά είναι γενικά πάρα πολύ σημαντικό το θέμα εν γέννη για την Επιτροπή μα. Ντομινίκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, τους ειδικούς για τις παρουσιάσεις που έκαναν. Έχω κάποια σχόλια, δύο σχόλια και μία ερώτηση. Το πρώτο σχόλιο. Στις διεθνείς διαδρομές, τις σιδηροδρομικές, ε, επιτρέπονται να γίνονται και μακρές διαδρομές. Εξεπλάγει από αυτά που είπε ο κύριος ε, Λόχμαν επί του θέματος. Μας εξηγεί ότι ε, υπάρχει ανταγωνισμός με τις εταιρείε χαμηλού κόστους αεροπορικές και τα κριτήρια της άνεσης πολυτέλειας ε, θα επέτρεπαν να επιβιώσουν τα νυχτερινά τρένα. Ε, η δυνατότητα να έχει εστιατόριο, να κάνει ντους κάποιος, να... όλα αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Η άνεση δίνει αυτά τα στοιχεία. Και εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τις ρεπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Προτείνεται διαφορετικός τρόπος μεταφορών. Λοιπόν, Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των τρένων και καμία στατική επιλογή που γίνεται μεταξύ του χαμηλού κόστους και των τρένων. Και α, είναι διαφορετική η νυχτερινή διαδρομή με τρένο που είναι άνετη. Μπορεί να υπάρχει ένα τρένο, νυχτερινό τρένο που να πλησιάζει πολύ τη μεταφορά ε, ζώων και μπορούμε να έχουμε νυχτερινά τρένα τα οποία είναι εξαιρετικά άνετα. Μπορείτε να διαλέξετε να μεταφέρει τους ανθρώπους μέσω των ε, τρένων που είναι άδεια την ημέρα, πιο γρήγορα την ημέρα ή πιο αργά το βράδυ. Λοιπόν, δεν είναι πολύ βανάγνωστη αυτή η διαφορά. Ε, δηλαδή, μπορεί κανείς να θέλει να μεταφέρεται, να ταξιδεύει αργά και άνετα και να διαλέγει το τρένο του. Μετά, η έκδοση εταιρείων ε, όσον αφορά τις μεταφορές είναι καταστροφική. Κανεί δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να ταξιδέψει απλά. Είναι πολύ περίπλοκο να δει κανεί μια προσφορά, να έχει μια προσφορά με ένα μόνο εισιτήριο σε διεθνή έκδοση εισιτηρίων. Η χρήση του διαδικτύου παραμένει εξαιρετικά πάρα πολύ προβληματική σε αυτό το τομέα. Τρίτον, η απόκτηση του, του ίδιου του εισιτηρίου, του χαρτιού, ε, ακόμα και του ηλεκτρονικού ε, εισιτηρίου είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Τέταρτον, υπάρχει η τιμολόγηση που είναι περίπλοκη. Ε, δυνατότητα μείωση, έκδοσης φοιτητών κλπ και τελικά δημιουργείται εντύπωση ότι ε, μπερδεύεται κανείς, σε, ε, μπερδεύεται κανείς όσον αφορά τους αριθμούς, ε, την τιμή κλπ. Λοιπόν, αναφέρεται ο συναγωνισμός με τις εταιρείε low cost. αλλά υπάρχει και το πρόβλημα να παχτήσει κανείς να βγάλει εισιτήριο χωρίς να απομακρύνεται από το σπίτι του. Λοιπόν, βλέπω ε, ότι υπάρχει κάποια αδιαφορία όσον αφορά το τρένο. Λοιπόν, μπορεί, ε, θα πρέπει να επεξεταστεί ε, η πολιτική που ακολουθείτε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι πραγματικές, υπάρχουν Όσον αφορά τιμολόγηση, χαμηλή τιμολόγηση, μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια, προβλέπετε κάτι για τον ανταγωνισμό με τις εταιρείες low cost. Βλέπω ότι η έλλειψη πολιτικής συντονισμένης μεταξύ των εταιριών στην Ευρώπη είναι τέτοια που δεν υπάρχει αξιόπιτη προσφορά από πλευράς πρακτικής προσέγγισης για τα τρένα και του ταξιδιού και από πλευράς άνεσης. Ευχαριστώ. Η Maya Κίλενεν ή ποιος? Α, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για αυτό το θέμα ανταγωνισμού μεταξύ τρένων και πούλμαν, λεωφορείων, έχει γίνει πολύ πιο επιθετικός. Έχουν ε, αρχίσει να λειτουργούν νέες εταιρείες πούλμαν που έχουν πολυτελή πούλμαν, χαμηλές τιμές. Έχει επηρεάσει αυτό τις ιδοδομικές μεταφορές. Και τι μέλλον βλέπετε, γιατί θα είναι σοβαρός ανταγωνιστής για το τρένο αυτές οι νέες εταιρείες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσει η Κομισιόν πώς θα προσπαθήσει να αναζωογονήσει, να εμψυχώσει τις σιδηροδρομικέ μεταφορές, γιατί ξέρουμε ότι μας λείπουν πολλά τμήματα συνδέσεων. Μας λείπουν νυχτερινέ γραμμές, μας λείπουν γραμμές σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Πρώτο αυτό. Ακούω αυτά που λέγονται, να θεωρήσουμε ότι πρέπει να είναι καλή η τιμή και ο χρόνος ε, μετάβασης δεν επαρκεί. Θεωρώ ότι σήμερα υπάρχουν προσφορές ε, που όλοι τη συγκρίνουν, ιδιαίτερα οι αεροπορικές εταιρείες ε, χαμηλού κόστους. Ορισμένοι αναφερθήκατε στα Πούλμαν. Τώρα ξέρετε γίνονται συνδυασμένες προσφορές, ε, λεωφορείο, συν Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές αυτές οι προσφορές πακέτου. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω. Να μάθω λέω τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε ε, να ξέρουμε και τι θέλουν σήμερα και τι θα θέλουν στο μέλλον οι επιβάτες. Μόνο με βάση τις ανάγκες τους μπορούμε να προσαρμόσουμε την προσφορά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρόεδρος. Πέτερ Λούντγκρεν. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ο χρόνος ε, είναι χρήμα. Εάν ε, πρέπει να κάνετε 12 ώρες με το τρένο ή 2 ώρες με το αεροπλάνο, είναι σαφές ότι θα προτιμήσετε την ταχύτερη επιλογή. Και πολλές φορές είναι και φθηνότερη πτήση. Αλλά υπάρχουν βέβαια μεγάλες ανησυχίες από πλευράς ανταγωνισμού. Διότι βεβαίως ε, χρειάζεται μεγάλη ανάγκη, χρειάζονται τρομερές υποδομές τρομερές επενδύσεις στις υποδομές. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους. Αλλά για να επιβιώσουν ε, οι σιδηρόδρομοι πρέπει να είναι φτηνά τα εισιτήρια. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει την συμμετοχή της ε, στους σιδηροδρόμους, αλλά δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Ξέρετε βέβαια όμως ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το τρένο. Το αεροπλάνο είναι ταχύτερο το αεροπλάνο. Και το θέμα είναι τι έχει στη διάθεσή του σήμερα ο επιβάτης. Οι επιβάτε, βέβαια μπορεί να θέλουν να μπορούν να κάνουν ντου στο τρένο, αλλά δεν είναι το κύριο να, αν θα μπορούν να κάνουν ντου. Το κύριο είναι να πάνε γρήγορα και φτηνά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να φτηνίνουν τα εστία των τρένων. Αυτό είναι το βασικό θέμα ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ζορς Μπαχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Διαπιστώνουμε ότι για διάφορες διαδρομές Υπάρχει προσφορά από διάφορες ε, εταιρείες που κάνουν ε, προσφορές ε, που λέγονται αλυσίδες, είναι αλυσιδωτές δηλαδή. Σκέφτεται η Κομισιόν εάν μια επιχείρηση θέλει να βγει από αυτήν την αλυσίδα για λόγους κερδοφορίας και επειδή αυτό θα οδηγήσει στην κατάργηση ολόκληρη αλυσίδα. Μπορεί η Κομισιόν να κάνει κάτι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, ανταγωνισμό με τι εταιρείε ε, χαμηλού κόστου. Εδώ συμφωνώ με τον ε, Ντομινίκ Ρίκε ότι πολύ σημαντικό είναι η ποιότητα του υλικού. Και διαπιστώνουμε ότι οι σιδηρόδρομοι έχουν επενδύσει πολύ σε υψηλού επίπεδου υψηλής ταχύτητας ε, βαγόνια και διαδρομές αλλά οι συμβατικοί σιδηρόδρομοι έχουν παραμεληθεί δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα να πληθείς ούτε δυνατότητα να πιείς έναν καφέ είναι πρόβλημα αυτό αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τις εταιρείε χαμηλού κόστους τότε πρέπει να είναι ανταγωνίσμη προσφορά μας σε αυτές τις συμβατικές γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρασκούν Μπιλμπάου τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω έτσι κάπως την εντύπωση ότι σε όλες τις συζητήσεις ε, μιλάμε για τα ίδια πράγματα, εστιάζοντας όμως κάπου διαφορετικά. Κάποια στιγμή πάντα ακούγεται στη συζήτηση το τέταρτο συνταδρομικό πακέτο, που δεν θα το καταλαβαίναμε ή δεν θα το ακούγαμε αν δεν είχαν ε, υποβληθεί προηγούμενες εκθέσεις. Τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ε, εισιτήριο και επειδή εγώ θέλω να αγοράσω από όπου θέλω το εισιτήριο και να πάω εκεί που θέλω χωρίς πρόβλημα, το να πάρω τρένο στο Στρασβούρο και να μην χρειάζεται να κατέβω σε μια άλλη χώρα πριν φτάσω στις Βρυξέλλες. Γιατί η Ευρώπη ε, συνεχίζει να έχει πάρα πολλά εμπόδια και δεν υπάρχει κανένα τρόπο να βελτιωθεί η κατάσταση, ούτε σε ό,τι αφορά την τιμή, ούτε στο να γίνει πιο ελκυστικό το τρένο για του ε, επιβάτε. Ούτε οι νυχτερινέ ε, γραμμέ ή τα ημερήσια τρένα ε, που είναι ελκυστικά. Άρα για το ίδιο πράγμα μιλάμε, αλλά βάζοντα αλλού την έμφαση κάθε φορά. Πρέπει όμως να ξέρουμε όλοι περί τίνο πρόκειται. Έχω μια ερώτηση προ τη Ομοσπονδία Δρόμων και μία προ την Ομοσπονδία των Επιβατών. Γιατί και οι δύο εκπρόσωποι ανέφεραν τη σημασία του να εγκρίνουμε τον τεχνικό πυλώνα από τετάρτου συνδρομικού πακέτου και να προχωρήσουμε. Όμω, αν δεν έχουμε τον, τον πολιτικό πυλώνα ή τη διακυβέρνηση, τι να κάνουμε τον τεχνικό πυλώνα. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μήπως πρέπει να είμαστε αντίθετοι με τα ιστορικά μονοπόλια και τις κυβερνήσεις και να προχωρήσουμε με ενίο τρόπο απέναντι σε αυτό το συνδρομικό πακέτο. Ακούλη τη μέρα αυτή τη συζήτηση και χθε και τον προηγούμενο και τον προ προηγούμενο μήνα. Και πάντα για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Όλα είναι γραμμένα. Βαρέθηκα, κουράστηκα να ακούω τις συζητήσεις αυτές. Έχουμε τη διάθεση να προχωρήσουμε. Με ειλικρίνεια όμως να το πούμε με τιμιότητα, με εντυμότητα. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν απέναντι σε αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να είστε και ειλικρινείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα εγγραφεί ο ίδιος ως τελευταίος. Με εντυπωσίασε 0,9% των οδών ε, έχουν διόδια και 100% των ε, σιδηροτροχιών. Καταστροφή αυτό. 6% του, των επιβατών του σιδηροδρόμου ε, διασχίζουν σύνορα. Θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών ε, που διασχίζουν σύνορα εδώ και 20 χρόνια και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Και τι κάνει η Κομισιόν. Είναι ανέντιμος ο ανταγωνισμός. Είναι τόσο φτηνές οι αεροπορικές εταιρείες, για, όχι επειδή τα πάνε καλύτερα, αλλά γιατί έχουν πάρει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια επιδοτήσεις. Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος κάθε χρόνο τους πληρώνει κάθε χρόνο 30 δις. Δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν πληρώνει για την κυροζήνη, ενώ οι σιδηρόδρομοι πρέπει να τα πληρώσουν όλοι. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβώς, ακριβά τα εισιτήρια του σιδηροδρόμου. Αυτά δεν προέκυψαν από τον ουρανό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και η Κομισιόν θα πρέπει να πει όχι, θέλουμε δίκιο ανταγωνισμό, όχι άδικο, πρέπει, όχι αθέμητο. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Η πώληση εισιτηρίων, η ενημέρωση για τα εισιτήρια, στο τρίτο πακέτο για τους αεροδρόμους, πριν από 7-8 χρόνια αποφασίσαμε τι πρέπει να γίνει. Και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Γιατί οι τιμές των εισιτηρίων για το διαμεθοριακό, για τις διαμεθοριακές σειροδρομικές μεταφορές τόσο διαφορετικές. Είμαστε ενωμένοι η Ευρώπη. Θέλουμε να υπάρχουν ενιαία εισιτήρια. Γιατί δεν υπάρχουν. Παράδειγμα, μεταξύ Βερολίνου και Μπρέσλα. Το ανάφερα ήδη. Μας λείπουν 50 χιλιόμετρα που θα μπορούσαμε να τα έχουμε με 100 εκατομμύρια και θα γλιτώναμε δύο ώρες. Ενώ τα υπεραστικά λεωφορεία, και όπως ξέρετε στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια, ενώ το υπεραστικό λεωφορείο κάνει 3,5 ώρες. Γι' αυτό σταματήσανε τη συνδρομική γραμμή γιατί είναι καλύτερο το λεωφορείο. Πριν από τον πόλεμο για αυτή τη διαδρομή το τρένο έπαιρνε 2,5 ώρες, τώρα παίρνει 5. Ε, πολλά, με 100 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή την τρύπα. Και τώρα σταμάτησε η γραμμή. Από την πλευρά της Πολωνίας μέχρι τα σύνορα, από το Βρότσλαβ λοιπόν μέχρι τα σύνορα, ε, είναι ηλεκτρική γραμμή. Αλλά από τα γερμανικά σύνορα μέχρι το Κότμπους, μόνο σε αυτό για αυτή τη διαδρομή είναι ηλεκτρική γραμμή. Και μετά υπάρχει αυτό το κενό. Και τι κάνει η Κομισιόν. Δίνει λεφτά για να σταματήσουν οι συνδρομικές μεταφορές. Καλά έχουμε τρελαθεί εντελώς. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Πού είναι η πρωτοβουλία της Κομισιόν να το αντιμετωπίσει αυτό, να το σταματήσει. Και για τα τρένα υψηλής ταχύτητας, το, το είπατε. Δεν είναι το σημαντικό η, η μέγιστη ταχύτητα, αλλά η μέση ταχύτητα. Έχουμε τον απολογισμό από το σύστημα TGV στη Γαλλία που από οικονομική πλευρά είναι καταστροφή. Και ακόμη και οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι λένε ότι αρκούν 250 χιλιόμετρα, όχι 350 γιατί τα πολύ ακριβά και επιβαρύνεται πολύ περισσότερο το δίκτυο. Τι επιπτώσεις ε, εξάγουμε. Πρέπει να κάνουμε πάντα τα ίδια λάθη. Πριν από 20 χρόνια αυτό που μας ενδιαφέρεται ήταν πάντα η μέγιστη ταχύτητα. Αλλά οι επιπτώσεις πρέπει επιτέλους, τα απορίσματα πρέπει επιτέλους να εξαχθούν, να αξιοποιηθούν. Πρέπει η Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό γιατί αλλιώ δεν έχει καμία δυνατότητα να επιβιώσει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και παρακαλώ τώρα να απαντήσετε σε όλα αυτά. Ποιο θα πάρει πρώτο το λόγο, ο κύριο Ζουνίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πράγματι συζητούμε πλέον το θέμα και η καρδιά του προβλήματος είναι ότι είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένοι οι σιδηρόδρομοι. Υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός μεταξύ της δυνατότητας σύνδεσης υπηρεσιών ε, από τη μια συνδρομικών και από την άλλη άλλων τρόπων μεταφοράς. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των συνδρομικών υπηρεσιών. Ανταγωνισμός, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερος δύσκολο. Είναι φορτισμένο ε, λόγω των διαφορετικών πλαισίων μεγάλη παράδοση. Έχουμε τη διαφορετική ιστορική παράδοση όλων αυτών των τρόπων μεταφοράς και είναι δύσκολο να βελτιωθεί η κατάσταση. Το γνωρίζετε όλοι αυτό. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Και αυτό όταν σας υποβάλλουμε νέες πρωτοβουλίες για την εσωτερική του εξωτερικού κόστους, που νομίζω ότι είναι η βάση που χρειαζόμαστε για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε πράγματι να λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις ε, και να προτείνουμε μέτρα για να μετατοπιστεί η ισορροπία ε, μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς να έχουμε μία εξισορρόπηση. Όμως πιστέψτε μας είναι δύσκολο και χρονοβόρο όλο αυτό. Δεύτερον, όποτε γίνεται λόγος για το σεδρομικό τομέα και χαίρομαι πολύ που πολλοί βουλευτές ε, ανέφεραν το τέταρτο σεδρομικό πακέτο, πράγματι εδώ προσπαθούμε με τις ενέργειές μας να βρούμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, ώστε οι νέες υπηρεσίες να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να είναι στο δυνατόν πιο προσβάσιμες, πιο ανοιχτές από ε, κυβερνητικής πλευράς, κρατικής πλευρά. Ελπίζουμε να υπάρχει πλήρης λογοδοσία με την υλοποίηση αυτού του πακέτου, να έχουμε τους διαχειριστές υποδομών που θα είναι ισχυροί και που θα διαβουλεύονται και θα συμπρογραμματίζουν, θα συνσχεδιάζουν και θα συνεργάζονται για να υπάρχει πανευρωπαϊκή έποψη και όχι μόνο εθνική έποψη των υποχρέσεων για επενδύσεις. Ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει σημαντικά πλεονεκτήματα. Άλλες πτυχές σίγουρα είναι σημαντική η ανοιχτή πρόσβαση. Αν κάνουμε παραλληλισμό είτε με τα λεωφορεία Πούλμαν ή τις πτήσεις, Είναι πολύ δύσκολο ακόμη στον τομέα των σιδηροδρόμων να ενσωματωθεί αυτό το δίκτυο. Υπάρχουν και ρυθμιστικά εμπόδια σε ό,τι αφορά τις τάσεις ε, στις ε, χώρες αγορές. Γι' αυτό χρειάζεται και μεγάλη βελτίωση για τις δυνατότητες που έχουμε. Η πρόταση PSO περιλαμβάνει αναφορά στη δυνατότητα ένα διεθνές ταξίδι μέρος του να καλύπτεται από αυτές τις υποχρεώσεις. Απαντώ σε μια από τις ερωτήσεις σας. Ο δημόσιος τομέας ε, χρειάζεται κάποιες φορές να παρέμβει για να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στους πολίτες. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις ε, τεχνικές πτυχές, η κυρία Μπιλμπάου και άλλοι πολύ καλά ανέφεραν τη σημασία όλες οι προτάσεις ε, να ενταχθούν στο τέταρτο συνδρομικό πακέτο γιατί ο τεχνικός πυλώνας πράγματι έχει ως στόχο την ε, μείωση του κόστους. Θέλουμε να έχουμε πιο οικονομικές υπηρεσίες και οικονομικά αγαθά. Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, συμφωνούμε με την απογοήτευσή σας και νομίζουμε ότι το πρώτο μέτρο που ελήφθη ήταν χάρη στον κύριο που είναι πίσω μου, ο κύριος Λίμπο Λόχμαν είναι υπεύθυνο. Θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και ο κύριος Λόχμαν και οι συνάδελφοι από την Κομισιόν υποχρέωσαν κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη, οπότε έχουμε πλέον συμφωνία τουλάχιστον για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Βέβαια, βραδέως κινούμαστε ακόμα, θα θέλαμε αυτό να το λύσουμε ε, σε συνεργασία με το σιδηροδρομικό τομέα, δηλαδή διευκόλυνσεις που υπάρχουν σε άλλες ε, μορφές μεταφορών να ισχύουν και για το σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες να μην είναι πιο ελεύθερα διαθέσιμες. Να μην μπορεί δηλαδή κανείς να κλείσει με διαφορετικούς τρόπους ε, το εισιτήριό του. Γιατί πρέπει μόνο να τα τυπώνει τα εισιτήρια σε ό,τι αφορά δε τη χρηματοδότηση των υποδομών. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί στις συνδρομικές προτάσεις που λαμβάνουμε, περισσότερες από τις προσπάθειές μας έχουν ως στόχο πράγματι να υπάρχει καλύτερη δυνατή συμμετοχή και των συνδρομικών σχεδίων. Κύριε Κράμερ, με τα νέα εργαλεία τα οποία μας έχετε παράσχει, βλέπουμε και τη διασυνοριακή σύνδεση, αυτή την πτυχή, ώστε με τις νέες επενδύσεις που έχουμε, παραδείγματος χάρη στη μία ε, πλευρά της μεθορίου να γίνονται και στην άλλη πλευρά και να μην έχουμε απομόνωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα ασχοληθώ με το τέταρτο πακέτο γιατί έγινε μία ερώτηση για τη γνώμη μας. Φυσικά για τις διεθνείς ε, υπηρεσίες επιβατών είναι ανοιχτές. Υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός εδώ και για το τέταρτο πακέτο, εμείς θα θέλαμε να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος για τον τεχνικό πυλώνα, γιατί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ε, μείωσης του κόστους. Όταν μιλάμε για διεθνείς υπηρεσίες επιβατών και για νυχτερινά δρομολόγια, αυτά θα παίξουν μεγάλο ρόλο για την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την ε, εξέλιξη των τεχνικών προδιαγραμμών, προδιαγραφών για την διαλειτουργικότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο τέτοιο σύστημα για τα βαγόνια επιβατών. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό το τμήμα των τεχνικών προδιαγραφών για να υπάρχει δυνατότητα αυτά τα βαγόνια να λειτουργούν παντού. Για τη διακυβέρνηση συμφωνώ. Χρειάζεται πλήρης διαφάνεια και οι διαχειριζόμενοι την υποδομή θα πρέπει να έχουν ε, κάθε ενημέρωση για το κόστος ε, πρόσβασης ε, στις τροχές. Αυτό λείπει ακόμη από τα προηγούμενα πακέτα των σειροδρομικών μεταφορών. Για τον ανταγωνισμό και την άρνηση παροχής υπηρεσίας και τις εταιρείε χαμηλού κόστους. Ναι, είναι ανώμια πράγματα αλλά είναι οι ίδιες αποστάσεις. Μιλάμε για αποστάσεις 800 με 1000 χιλιόμετρων. Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός. Φυσικά, αν πάρω αεροπλάνο για μια μισή ώρα, δεν θα ήθελα πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Αλλά αν πρέπει να πάρω το τρένο 8-10 ώρες, τότε απαιτώ, περιμένω ένα κάποιο επίπεδο. Άρα τα τρένα πρέπει να προσφέρουν οπωσδήποτε πολύ υψηλότερη ποιότητα. Και αυτή η ποιότητα όμως ε, αντανακλάται και στην τιμή του εισιτηρίου. Και το κόστος έχει να κάνει και με τα τέλη και την ε, συμμετοχή ε, του εξωτερικού κόστους στην τιμή του εισιτηρίου. Και ελπίζω όταν θα μιλήσετε για τα διόδια τα απόγευμα και τα τέλη στο μέλλον, να βάλετε αυτό το στοιχείο. Πώς συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο το συνολικό κόστος των υποδομών. Αυτό θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό για τους σιδηροδρόμους. Εισιτήρια, βεβαίως, μπορούμε να βελτιώσουμε την τιμολόγηση. Το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό έχουμε αυτό το πρότυπο πλήρους υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι ε, η κοινή δυνατότητα να μπορούν να αγοράσουν όλες τις υπηρεσίες επιβάτες και αεροπορικές και σιδηροδρομικές. Δηλαδή τα εισιτήρια πρέπει να αφορούν και όλους τους τρόπους μεταφοράς. Φυσικά δεν θα έχουμε βελτιώσεις για τους επιβάτες από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρξει και η αλλαγή του λογισμικού. Αλλά οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα. Ανταγωνισμός τρένου και λεωφορείων. Παρατηρούμε ότι όπου έχουν ε, εισαχθεί στο δίκτυο αυτά τα λεωφορεία έχουν πάρει μερίδιο της αγοράς από τα τρένα, διότι και τα λεωφορεία όπως και τα αεροπλάνα είναι πολύ φθηνότερα. Γιατί έχουν ε, χαμηλότερο κόστος ε, λειτουργίας. Ιδού λοιπόν ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέλλον των διεθνών σιδεροδρομικών μεταφορών επιβατών. Και αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στα νυχτερινά δρομολόγια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ρίλα Γκέροντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία-τέσσερα πράγματα θέλω να πω. Ας ξεκινήσουμε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Όπως και οι συνάδελφοί μας, οι φίλοι μας στο CER και εμείς θέλουμε να δούμε τον τεχνικό πυλώνα να γίνει νόμος. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, υποστηρίζουμε την αρχή της φιλελευθεροποίησης αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι οι σιδηρόδρομοι να εξακολουθούν να λειτουργούν ως ομάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μεγάλο κατακαιρματισμό των δικτύων κατακαιρματισμό της προσφοράς προς τους επιβάτες. Όσο πιο μεγάλο το ταξίδι, το διεθνές που κάνει κανείς, μιλάμε βασικά για διεθνή ταξίδια, πιο πιθανό είναι να είναι πολυτροπικό ταξίδι. Άλλο παράδειγμα. Ανέφερα το νυχτερινό τρένο πριν από δύο εβδομάδες που πήγα από το Άμστερνταμ στο Μόναχο. Ήταν ένα κομμάτι πολυτροπικού ταξιδιού, ξεκίνησε στην πόλη μου στην Ανατολική Αγγλία, 40 λεπτά σε τρένο, 20 λεπτά ταξί, πτήση πάνω τη Βόρεια Θάλασσα, 50 λεπτά περίπου, τοπικό τρένο από το Σίπολ, το αεροδρόμιο προς το κέντρο του νυχτερινό ταξίδι στο Μόναχο, ημερήσιο τρένο διεθνές, Μόναχο Σάλτσπουργκ και μετά ποδαρόδρομος για τα τελευταία δεκά λεπτά. Αυτό ήταν το ταξίδι μου, πόρτα σε πόρτα. Χρειάζεται πολυτροπική λειτουργία πρόσκοπτη να αναφερθώ στα λεωφορεία και στις ε, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Έχω χρησιμοποιήσει πτήση χαμηλού κόστους το φθινόπωρο, Λονδίνο-Βουκουρέστι. Και για να πω ειλικρινά, βασικά λόγω κόστους και χρόνου. Θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερο χρόνο να πάω σιδηροδρομικός και θα κόστιζε περισσότερο. Στην Αγγλία λέμε ότι διαλέγεις το πιο συγκεκριμένο τρόπο που σε βολεύει το ταξίδι σου. Και καμιά φορά και για την τσέπη σου. Για το εισόδημά σου. Οπότε έρχομαι στο αρχικό μου σημείο. Δηλαδή οι διεθνείς επιβάτες πρέπει να έχουν λογική δυνατότητα επιλογής και θα πρέπει ισότιμα να παρέχεται μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς οι επιλογές. Μετά τα βαγόνια για τα διαδρομές, μα, συγγνώμη, τα υπεραστικά πούλμαν, λεωφορεία. Τα χρησιμοποιούν κάποιοι για κάποιους λόγους. Πρώτα απ' όλα λόγω κόστους. Δεύτερον, διότι ένα ταξίδι με λεωφορείο ίσως να είναι απλούστερο από ότι με τρένο. Κυρίως αν συνδέει δύο μέρη όπου δίδυ συνδέονται εύκολα σιδηροδρομικά. Οπότε καμιά φορά εξετάζει κανείς τον δεχόμενο εναλλακτική λύσεω. Μήπως μπορώ να πάω μέσω πούλμαν αντί να πάω με τρένο. Τούτου λεχθέντος είναι ζωτική σημασία να χρησιμοποιεί τα σωστά τερματικά το λεωφορείο, να μην σε αφήνει ξημερώματα σε κάποιο σκοτεινό δρόμο, όπως κάνουν κάποια λεωφορεία, και να υπάρχει συγκρίσιμο επίπεδο φροντίδας για τον επιβάτη και ενημέρωση με τα τρένα. Άρα μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, αλλά σε κάποιο βαθμό αυτός ο ρόλος έχει σχεδόν, διαδραματίζεται σχεδόν αυτόματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο και ακούσαμε τις παρουσιάσεις. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας να κάνουμε, αλλά ευχαριστώ τον κύριο Ουνίδη που ανήγγειλε ότι θα εργαστεί για να συμπεριληφθεί στο εισιτήριο το κόστος το συνολικό κόστος. Πρέπει να συμβεί αυτό. Για παράδειγμα, γιατί ενώ τα αεροπλάνα δεν πληρώνουν φόρο για την κυροζήνη τους, πληρώνουν για το καύσιμό τους τα τρένα. Ενώ για τις διεθνείς πτήσεις δεν υπάρχει ΦΠΑ, για τα τρένα υπάρχει. Αυτά θα πρέπει να το πούμε στα κράτη-μέλη. Να επιβληθεί ΦΠΑ. Ισότητα δικαιωμάτων. Καλό θα ήταν. Σας υποστηρίζουμε Παρακαλώ να μας κάνετε σύντομα προτάσεις. Βέβαια, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά όχι και πολύ αργά. Επόμενο θέμα. Πριν περάσω σε αυτό, να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από την κάτω Σαξονία που μόλις κάθισε. Καλώς ήρθατε παρακαλώ στην Επιτροπή μας. Τους έχει, ε, ε, ε, είναι προσκεκλημένη της κυρίας Μάσινα. Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση ε, Έχουμε μία έκθεση για τον οργανισμό για τη θαλάσσια ασφάλεια. Καλώς ήρθατε. Κύριε Μίλη, σας δίνω το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ και μου δώσατε τη δυνατότητα να σας πω λίγα λόγια για τις τρέχουσες δραστηριότητες ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και για το ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας η οποία πάντοτε μας στήριζε και ήταν και πολύ σημαντική για όλη την πορεία μας από τότε που ιδρυθήκαμε το 2002. Είχα κάνει και μια πρώτη παρουσίαση το 2012 ο πρόεδρος. Παρακαλώ σιωπή, ησυχία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τακτή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής σας και του οργανισμού μας και γι' αυτό θέλω και εγώ να παραμείνει ανοιχτός αυτό ο διάβολο, επικοινωνία και στο μέλλον. Όπως ε, ε, γνωρίζουμε είστε ε, πολλοί από εσάς νέοι βουλευτές. Θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω τον οργανισμό μας, το προσωπικό, τι υπηρεσίες προσφέρουμε και θα πω και λίγα λόγια για την πενταετή στρατηγική που πριν από λίγο καιρό υιοθετήσαμε. Ο οργανισμό μα είναι ένα από του εκτελεστικού οργανισμού που δημιουργήθηκαν το 2002 μετά την ε, έγκριση ειδική ε, τεχνική νομοθεσία στον τομέα τη ε, θαλάσσιας ασφάλεια, Μιλώ για τη δέσμη μέτρων ΕΡΙΚΑ 1 και 2. Ως εκτελεστικό οργανισμό, έχουμε εντολή την εντολή αυτή την ορίζει ο κανονισμός, ο, κανονισμός του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε νομική προσωπικότητα, προϋπολογισμό και Είμαστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητές μας. Από το 2006 έχουμε έδρα τη Λισαβόνα. Πριν από πέντε χρόνια εγκαινιάσαμε τα κεντρικά μας γραφεία εκεί και είμαι υπερήφανος γιατί διευθύνω το κέντρο αριστείας αυτό με 250 άτομα προσωπικό όλη την Ευρώπη. Ε, εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γέννη την ε, ναυτιλιακή δέσμη, το ναυτιλιακό κλάστερ. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. 55 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι ο προπολογισμό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έσοδά μας είναι γύρω στα 400.000 έσοδα το χρόνο μόλις ε, και 1,5 εκατομμύρια είναι η συνεισφορά της ε, ΕΖΕΣ, της ΕΦΤΑ. Ε, όταν είχα έρθει στην Επιτροπή σας το Σεπτέμβριο του 2012, Είχαμε την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού μας, του ιδρυτικού κανονισμού, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Άρχισε να ισχύει από το Μάρτιο του 2013 και κάνει τη διάκριση μεταξύ των βασικών και των επικουρικών ε, καθηκόντων μας. Υπάρχουν ε, τα βασικά καθήκοντα που παραμένουν, αλλά έχει πλέον ε, διευρυνθεί το πεδίο των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων γιατί πλέον συμπεριληφθήσαν οι καταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχουμε επίσης σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια επιτήρηση, η τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στους εταίρους μας από τις πολιτικές γειτονίες έχει διευρυνθεί. Όμως δεν είμαστε εξαίρεση σε σχέση με άλλους εκτελεστικούς οργανισμούς. Μας ζητήθηκε λοιπόν να μειώσουμε και το εργατικό μας δυναμικό και το προπολογισμό μας για τα επόμενα χρόνια. Άρα, πρόκλησή μας είναι να ε, έχουμε μεν αυτές τις περικοπές, χωρίς όμως αυτό να είναι σε βάρος ε, των πετικών μας υπηρεσιών. Πρόσφατα εγκρίναμε τη νέα πενταετή στρατηγική του οργανισμού μας, ε, την οποία και εκπώνησα σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το έργο του οργανισμού μας για την επόμενη πενταετία με βάση ύψες της σημασίας αρχές, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ευελιξία και δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Βασιζόμαστε στο όραμα ότι είναι όριμο αρκετά πλέον ε, το όργανο αυτό για να παρέχει ποιοτικέ υπηρεσίες, ιδίως στους βασικούς ε, διαφερομένους φορείς, αλλά και γενικότερα στον τομέα της ναυπηλίας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία και θα σας πω μετά και ποια είναι η δική μου έποψη και το δικό μου όραμα για την επόμενη πενταετία. Κάνουμε πολύ σημαντική δουλειά ε, υποστηρίζοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης ε, των ε, νομικών πράξεων. Κάθε θαλάσσια διοίκηση σήμερα πρέπει να εφαρμόσει μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οποίες έχετε συνεισφέρει και εσείς ως Επιτροπή. Πρόκειται για νομοθεσία η οποία θέτει πολύ ψηλά ποιοτικά πρότυπα. Είναι λοιπόν ε, οι λιμένες ε, και οι ευρωπαϊκές σημαίες ε, σύμβολα ποιότητας και θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη ομοιόμορφα ενιαία να τηρούν την νομοθεσία και Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τακτικές επιθεωρήσεις ε, και επισκέψεις και δίνουμε τους ελέγχους αυτούς ε, και τα πόρισματα στις υπηρεσίες της Κομισιόν. Επίσης θέλουμε οι επιθεωρητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ελέγχουμε τα περιφερειακά, τα γραφεία και κάνουμε και επισκέψεις ώστε και οι εταιρείε νεολόγησης να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά όταν επιθεωρούν την οπίγηση νέων πλοίων ή την επισκευή παλαιότερων. Επίσης, ε, για να δώσω ένα παράδειγμα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούμε την πρόσφατη συγχώνευση του DNV Νόρς και Βέριτας ε, και της ε, γερμανικής Λόιτ, που είναι δύο εταιρείε νεολόγησης, γιατί έχουμε ως στόχο τη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων Μπορεί να γνωρίζετε ότι πολλές ακτοπλοκές εταιρείες εκτός ε, Ευρώπης εργάζονται ε, σε πλοία με ευρωπαϊκή σημαία. Το σύστημα που έχουμε στη διάθεσή μας προβλέπει η Κομισιόν και ο οργανισμός μας να επιθεωρεί τα συστήματα, ε, μεταξύ άλλων και τα συστήματα πιστοποίηση εκ μέρου των κρατών μελών. Υπάρχει μια κοινή μεθοδολογία και έτσι εξοικονομούμε πόρου από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Και ταυτόχρονα έχουμε μια ε, ομοιογενή προσέγγιση. Παράδειγμα, πολλοί, έρχονται από τις, ε, πολλοί ναυτικοί προέρχονται από τι Φιλιππίνε, για παράδειγμα. Και υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα ελέγχων για να βεβαιωθούμε ότι τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις οι Φιλιππίνες. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον αρκετή οριμότητα για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο μέλλον. Έχουμε μια προσέγγιση στις ελέγχους μας που βασίζεται στην ελέγχη των κινδύνων. Έχουμε ένα κύκλο ελέγχων και διάδοση των αποτελεσμάτων, των οριζόντιων αναλύσεων και ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών. Ο οργανισμός μας επίσης δραστηριοποιήθηκε στην υλοποίηση ορισμένων καθηκόντων στον τομέα της περιβαλλοντικής ε, θαλάσσιας προστασίας, ε, παρέχοντας ε, αρρωγή στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τα πλοία. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε και ελέγχουμε σε διεθνές επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΕΜΣΑ εξεργάζεται την οδηγία το, την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων και έχουμε αναπτύξει μια σειρά εγχειριδίων, οδηγιών για τη δημοτοληψία, την αναφορά κτλ. Και επίσης αναπτύξαμε ένα ειδικό σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επιθεωρήσεις ότι αφορά το θείο μεταξύ των αρμοδιών και των διοικήσεων. Πρόκειται για ένα έργο που συνεχίζεται και με άλλους τρόπους ε, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις οδηγίας. Τεχνική στήριξη για τη χρησιμοποίηση του υγραερίου και τα λοιπά. Για τα επόμενα χρόνια θα ήθελα ε, ο ΕΜΣΑ να εστιάσει την εμπειρογνωμοσύνη του για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την πρόληψη της, ε, ε της ρήπανσης με την παροχή τεχνικής συνδρομής στους ενδιαφερόμενους φορείς και βέβαια ε, ένα ενδεχόμενο είναι και η δυνατότητα χρήσης των ε, συστημάτων πληροφοριών. Επίσης, υπάρχουν ε, εθνικά συστήματα προηγμένα συστήματα πληροφοριών για τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, για παράδειγμα. Έχουμε αναπτύξει και συντηρούμε ένα σύστημα ανταλλαγής θαλάσσιων πληροφοριών, SafeSynet λέγεται. Εδώ συνδυάζουμε όλα τα εθνικά συστήματα σε ένα ευρωπαϊκό και υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Κάθε ε, διαπιστευμένος χρήστης του συστήματος μπορεί να τις αποκτήσει απλά κάνοντας ένα κλικ σε οποιαδήποτε από αυτά τα τρίγωνα. Καθένα αυτά αντιστοιχεί σε ένα πλοίο. Εδώ βλέπετε ένα στιγμιότυπο ε, στο, στο φυσικαϊκό κόλπο ε, για μια συγκεκριμένη ημέρα ή ώρα. Και έχουμε έκθεση για 5 εκατομμύρια θέσεις. Και 5.000 διαφορετικές ε, κοινοποιήσεις ε, για τις θέσεις, ε, τα τα κτλ. Τελευταία εχμή της τεχνολογίας είναι να χρησιμοποιούμε και τη δορυφορική τεχνολογία. Έχουμε λοιπόν το δορυφορικό προηγμένο σύστημα πληροφοριών για την, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πλοίων. Έχουμε επίσης και το ELRI, το σύστημα αναγνώρισης εξαποστάσεως παρακολούθησης πλοίων Παρακολουθούμε όλο αυτό το σύστημα με δορυφορική πλοήγηση και επικοινωνία. Με, τις εικόνες αυτή με την εικόνα αυτή βλέπετε πάλι τον ίδιο ε, κόλπο, αλλά αυτή τη φορά στο πλαίσιο του LRIT. Χάρη στην ευέλικτη αρχιτεκτονική των υπηρεσιών μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες σήμερα από όλους, όλες τις θαλάσσιες ναυτιλικές εφαρμογές. Και αυτό μας δίνει μια πολύ πληρέστερη και ορθότερη εικόνα. Γιατί ο συνδεσμός πολλών συστημάτων μπορεί να ευνοήσει την εσωτερική αγορά και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών. Ένα άλλο παράδειγμα για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ολοκληρωμένου συστήματος και τη συλλογή πληροφοριών και παροχής όλων των πληροφοριών ήταν η πρόσφατη επιδημία του ιού έμπολα. Καταφέραμε να δώσουμε πληροφορίες για τα πλοία που είχαν καταλήψει χώρες ε, ε, που είχαμε κρούσματα του ιού και τα οποία έπλεαν ε, στα ευρωπαϊκά ύδατα ή πλησίαζαν τα ευρωπαϊκά ύδατα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη για να έχουν στοχευμένα μέτρα. Ο εντοπισμός πλοίων δεν είναι η μόνη δυνατότητα που μας δίνουν οι εξέλιξεις της δορυφόρικης τεχνολογίας. Ε, μπορούμε και κάποιες λεγόμενες επιχειρησιακές ε, πετρελοκυλίδες να τις εντοπίζουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πλοία τα οποία περνούν ε, το βράδυ κυρίως κάνουν τον καθαρισμό των δεξαμενών και έχουμε εκατοντάδες κοιλίδες τέτοιες που μπορούμε να εντοπίσουμε χάρη στη συνεργασία μας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Όταν λοιπόν ο δορυφόρος εντοπίσει μια πτρελοκυλίδα, το παράκτιο κράτος που είναι αρμόδιο για αυτή την περιοχή λαμβάνει ένα ε, προειδοποιητικό μήνυμα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να στείλει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της κυλίδας και να λάβει τις απαιτούμενες δράσεις ε, για την απορρίπανση. Επίσης, αυτό έχει και ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα, γιατί πολλές παράνομες ε, κροές ε, μειώνονται και μάλιστα δραματικά σε σχέση με το παρελθόν. Αλλάζει το τοπίο γρήγορα και η ΕΜΣΑ έχει αναπτύξει τις δυνατότητες της για τη συλλογή και ενσωμάτωση στοιχείων από οποιοδήποτε σύστημα του οργανισμού και από εξωτερικές πηγές, ούτως ώστε να είναι πληρέστερη εικόνα των τεκτενομένων στη θάλασσα αυτό με τη σειρά του μπορεί να προσαρμοστεί ιδεόντως και να ανακατεμηθούν οι πληροφορίες σε κράτη μέσα Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε άλλους φορείς. Οπότε το χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων αυξάνεται. Αναλύεται καλύτερα η κατάσταση στις θάλασσες ε, σε κάθε στιγμή. Αυτό ισχύει για τη Frontex που δέχεται από την ΕΜΣΑ πληροφορίες σχετικά με τις θάλασσες για το σύστημα, το Eurosur που είναι για την εποπτεία των συνόρων και αφορά τον έλεγχο και εντοπισμό των σκαφών. Παρέχουμε πληροφορίες και στην Υπηρεσία Ελέγχου της Αλληλείας, την ΕΦΚΑ, που ελέγχει την παράνομη αλληλεία. Επίσης συμβάλλουμε στην UNAFOR όταν προσπαθούν να καταπολεμήσουν ε, ε, την πειρατεία στο κέρας Αφρικής. Στο μέλλον θέλω ο οργανισμός να παγιώσει το ρόλο του ε, σαν πάροχο ε, δεδομένων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι θαλάσσιε δραστηριότητε. Πρέπει να αποκτήσουμε και νέε δυνατότητε λόγω τη ε, τεχνολογία στον έλεγχο των θαλασσών και να διερευνήσουμε τον τρόπο υποστήριξη άλλων κοινοτήτων παρέχοντας αξιόπιστα στοιχεία, αποφεύγοντας όμως και αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών. Ο οργανισμός επίσης έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά την αντίδραση στις στη ρήπανση μετρολογική λίδε. Ε, έχουμε 18 σκάφη για την απορρίπανση στις ακτέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Έχουμε 2 σκάφη στη Βαλτική, 3 στη Βόρεια Θάλασσα, 4 στη, στην ακτή του Δυτικού Ατλαντικού, 6 στη Μεσόγειο και 2 στον Εύξηνο Πόντο. Λειτουργούν ε, με σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα αυτά τα σκάφη. Εμείς καθορίζουμε τις προδιαγραφές για την αντίδραση στη ρήπανση και παρέχουμε και τον εξοπλισμό. Τα σκάφη ε, λειτουργούν μέσω ιδιωτών πλειοκτητών που ασκούν δική τους εμπορική δραστηριότητα στις θαλάσσιες περιοχές αλλά που έχουν υπογράψει μια συμφωνία ετοιμότητας, σύμβαση ετοιμότητας με την ΕΜΣΑ. Δηλαδή αμέσως θα σταματήσουν την εμπορική τους δραστηριότητα και θα κινηθούν προς δραστηριότητες απορρίπανση σε περίπτωση μεγάλου προβλήματος πρέπει να είναι έτοιμοι για αντίδραση έναντι της ρήπανσης σε 24 ώρες. Ε, είχαμε και την έκρηξη στην ε, μονάδα ε, εξόριξης πετρελαίου στην, στον κόλπο του Μεξικού. Έχουμε πάνω από χίλιες εγκαταστάσεις για το αέριο και το πετρέλαιο στην Ευρώπη και αυτές οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε ρηχά ύδατα που έχουν βάθος λιγότερο των 300 μέτρων όπως ανέφερα η δυνατότητα μας αντίδρασης στις πετρελοκυπηδίδες θα πρέπει να αντιδράσει δεόντω, δεόντως λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο. Διότι τώρα συμπεριλαμβάνουμε και τη ρήπανση και από τις μονάδες εξόριξης πετρελαίου της θαλάσσιας. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε πετρελοκυλίδα από πλοίο και από μονάδα εξόρυξης ε, η πετρελοκυλίδα διαφέρει σε φύση και τοποθέτηση θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή υπηρεσία για ενέργεια καταπολέμηση των κυλίδων και να υπάρχει δυνατότητα ψεκασμού. Εκεί έχουμε κάποιο κενό και πρέπει προσπαθούμε να το καλύψουμε. Θέλουμε να εξοπλίσουμε και τα πλοία ε, ανάκτησης με συστήματα ψεκασμού ε, παρόλο που εμείς προτιμούμε να έχουμε μηχανικά συστήματα απορρίπανσης. Ε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι αυτή η σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων σας έδωσε κάποια γεύση του τι κάνουμε στον οργανισμό μας. Επίσης προσβλέπω στις ερωτήσεις σας και θα ήθελα να σας ε, πω ότι η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή στην ΕΜΣΑ. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον οργανισμό μας στη Λισαβόνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μίλη. Είστε διευθυντής ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσια Ασφάλειας και νομίζω ότι το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους ε, προσκεκλημένους μας από την κάτω Σαξονία που έχει μια πολύ εκτεταμένη ακτογραμμή. Δεν θα ακολουθήσουμε τώρα τη σειρά των συντονιστών. Όποιος θέλει το λόγο μπορεί να τον πάρει. Πρώτη είναι η Deirdre Κλούν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που σχημάτισε μια πολύ καλή εικόνα για τις υπηρεσίες που παρέχετε και που στηρίζεται τα κράτη-μέλη. Ερώτηση συγκεκριμένη. Αναφερθήκατε στους ναυτικούς και τους Φιλιππινέζους. Ήμουν σε μια διάσκεψη για αυτό το θέμα πρόσφατα και αναφέρθηκε το θέμα προσέλκυσης ατόμων εργαστούν στον τομέα της ναυτιλίας που είναι κάτι προβληματικό. Δεν θεωρείται σαν καριέρα ε, που μπορεί να προδέψει κανείς δεν είναι ελκυστική. Και για την οικογενειακή ζωή δεν είναι ελκυστική η ζωή του ναυτικού. Σε ποιο βαθμό είναι πρόβλημα αυτό. Πολλά που αναφέρατε τα προβλήματα εξαρτώνται από τεχνογνωσία του πληρώματος. Υπάρχουν πολλά πλοία στα ύδατά μας. Έχετε κάποια στοιχεία. Σε ποιο βαθμό είναι πρόβλημα όσον αφορά τις αμοιβέ που μπορούν να προσελκύουν ναυτικούς. Και δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των γυναικών. δεν τραβάει τις γυναίκες στο επάγγελμα του ναυτικού. Είναι πρόβλημα και γίνεται πιο εμφανές όσο συνομιλώ με ανθρώπους ε, του τομέα. Γκεζίνε Μάισλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μίλη για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ε, είμαι από την κάτω Σαξονία που έχει τόσο εκτεταμένη ακτογραμμή, παρόλα αυτά ενδιαφέρομαι. Πολλά σχόλια θα είχα, θα περιοριστώ σε ορισμένα. Έχουμε την στρατηγική για την ε, γαλάζια ανάπτυξη. Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο οργανισμός σας σε αυτό. Έχω κάποιες αντιλήψεις, αλλά θέλω τη δική σας αντίληψη. Διότι η γαλάζια ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό για να δημιουργηθούν και θέσει εργασία. Δεύτερον, πολύ καλό που μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου είστε υπεύθυνο και για την ε, έρευνα και τους ελέγχους για τις πετρελαιοκυλίδες. Ξέρουμε ότι είστε υπεύθυνοι γι' αυτό και από τα πλοία και από τις πλατφόρμες. Πολύ καλό αυτό. Τρίτον, Είπατε ότι έχετε ένα δίκτυο για τη συλλογή στοιχείων και μέσω των δορυφόρων. Οπότε η ερώτησή μου, έχετε όλα τα στοιχεία που θα χρειάζεσταν, θα χρειαζόσασταν και για τον τομέα της αλληλείας για παράδειγμα. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές ε, δεν μπορούμε να λάβουμε τέτοια στοιχεία από τα κράτη-μέλη ή από άλλους που παίζουν ρόλο. Έχετε λοιπόν μια δυνατότητα πλήρους ε, και πώς εγγυάστε την προστασία των δεδομένων, να μην γίνεται κατάχρησή τους. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να μπορούμε να συλλέγουμε αλλά και να προστατεύουμε τα στοιχεία. Κάτι ακόμη. Ξέρω ότι για το θέμα του ιού έμπολα ε, ε, παίζει μεγάλο ρόλο η προστασία στα αεροδρόμια. Τι πρακτικές επιπτώσεις έχει αυτό, αν ξέρετε ότι κάποιο πλοίο έρχεται από περιοχή έμπολα, τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει όλο το πλήρωμα να μπει σε καραντίνα. Υπάρχει κάποια, κάποιο κρούσμα έμπολα μέσω των θαλασσίων μεταφορών. Βέβαια η περίπτωση του Φλαμίνια, αυτού του σκάφους από την, Άτο από την κάτω Σαξονία που υπέστη κάποια βλάβη και που κανείς ε, δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη. Τι πορίσματα εξάγεται δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να μπορούμε να δράσουμε καλύτερα. Και κάτι ακόμη. Σε τι βαθμό θα βοηθούσε αν θα μπορούσαμε όλοι να ε, μιλάμε μόνο αγγλικά στον τομέα των θαλασσιών μεταφορών. Ευχαριστώ. Κύριε Κίθ Taylor, μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά. Ήξερα ότι υπήρχε κάπου ένα κουμπί, το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Το θέμα είναι οι συμπροματικές ευθύνες που ανέθεσε στην έμψα το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις ε, πλατφόρμες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ήμουνα εισηγητής για την νομοθεσία, για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση για αυτές τις ευθύνες. Για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο αυξήθηκε ο βασικός προϋπολογισμός για την ΕΜΣΑ κατά 165 εκατομμύρια ευρώ στην περίοδο αυτή. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας ενημερώσετε σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΜΣΑ όσον αφορά τις, ε, τις παρακολουθείς στην εποπτεία των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχετε κάποια σχόλια χρήσιμα όσον αφορά την οικονομική στήριξη που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι που θέτω εκ νέου ένα ερώτημα, αλλά κύριε Διευθυντά, μπορείτε να μας πείτε τίποτα για την συνεργασία με τους εθνικούς φορείς να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, να μην είναι πολύ δαπανηρή η δραστηριότητα και να μην υπάρχει επικάλυψη από την άλλη στο έργο που επιτελείται. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια απάντηση πάνω σε αυτό. Μπορείτε να μας πείτε πώς συνεργάζεστε με τους εθνικούς φορείς, κυρίως για να αποφευθούν αλληλεπικαλύψεις. Ως εφαρία. Καλημέρα. Κύριε Μάρκο Μίλε, σας συνάντησα στην ΕΜΣΑ στη Λισαβόνα με τα χαράς. Όλες οι ερωτήσεις ε, που έθεσα ήδη απαντήθηκαν. Δεν έχω ερώτηση. Να σας πω όμως ότι η παρουσίασή σας όχι μόνο εδώ, αλλά η όλη παρουσίασή σας που μου κάνατε στην Λισαβόνα ήταν υπέροχη. Και η βάση δεδομένων της ΕΜΣΑ είναι εντυπωσιακή. Νομίζω ότι όλοι έπρεπε να επισκεφθούν στη Λισαβόνα την ΕΜΣΑ να δουν επιτόπου την παρουσίαση της ΕΜΣΑ. Θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι το παράδειγμα που δώσατε για τον ιό του έμπολα είναι ένα μικρό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ΕΜΣΑ για, την, ε, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσον αφορά τη συλλογή και διαβίβαση των διαθεσίμων στοιχείων. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανε τα τελευταία χρόνια η ΕΜΣΑ και πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Οπότε παρακαλώ απαντήστε και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. υπάρχουν ατυχήματα. Και όταν υπάρχουν ατυχήματα θα πρέπει το πλοίο να μπορεί να πάει στο πλησιέστερο λιμάνι. Γίνονται όμως πάντα ε, μεγάλες συζητήσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη, ούτε με την ασφάλεια μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που συνέβη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που δεν μπόρεσε να πάει στο πλησιέστερο λιμάνι. Τι πρέπει να κάνουμε, όλοι πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά κανείς δεν τα κάνει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με τους ναυτικούς και τα κοινωνικά μέτρα. Τι μπορεί να κάνει η ΕΜΣΑ για να προσελκύσει ναυτικούς. Το συζητήσαμε εδώ και μια εβδομάδα στη συνάντηση των διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θαλάσσια θέματα και προβληματίζονται όλα τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Διότι μειώνεται ο αριθμός των ναυτικών στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να το εξετάσουν και η ΕΜΣΑ. Αν δει κανείς το έργο που επιτελείται στα σκάφη, ε, αυτό είναι κάτι που δεν προσελκύει πολύ τους νέους να γίνουν ναυτικοί. Παρόλο που είναι σύγχρονα τα σκάφη, έχουν εξοπλιστεί με υψηλή τεχνολογία και πρέπει να το πούμε στους νέους ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτούς στα σκάφη με τις νέες τεχνολογίες και έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν ε, τις σπουδέ τους ε, και μετά την καριέρα τους στη θάλασσα. Μπορούν να βρουν και μετά δουλειές στη στεριά μετά την εμπειρία που αποκομίζουν. Είναι δύσκολο έργο για μας. Όπως σας ανέφερα, Έχουμε 70 με 75% των σκαφών με ευρωπαϊκή σημαία που χρησιμοποιούν ναυτικούς από την Άπο Ανατολή. Από πλευρά αμοιβών να πω ότι η στα σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία για τα πληρώματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω είναι αρκετά ελκυστική. Οι ναυτικοί από τρίτε χώρες βέβαια πληρώνονται λιγότερα, αλλά όλο και περισσότεροι ναυτικοί προέρχονται από τρίτες χώρες για την ώρα. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και ο IMO επίσης το ανέφερε αυτό και το τόνισε τα τελευταία χρόνια. Τι έκανε η ΕΜΣΑ για να ε, υποστηρίξει ε, την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δώσαμε πολλές πληροφορίες για να ελέγξουμε να ελέγξουμε διοικητικά τα σκάφη για την γαλάζια ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε προσπάθειες το 2010-2011, μελετήσαμε τις δυνατότητες που υπήρχαν για να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό άχθος επί των σκαφών με τέτοια βαθμολόγηση στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είχαμε 250 σκάφη που παρακολουθούμε και παρακολουθήσαμε τακτικά και με τα συστήματά μας μπορούμε να παρακολουθούμε τα σκάφη και να χρησιμοποιούμε τα συστήματά μας ούτως ώστε οι αρχές να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για σκοπούς φορολόγησης. Βασικό εμπόδιο είναι ότι οι αρχές, οι εφορίες δεν δέχονται τις ηλεκτρονικές μεθόδους α, πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι αυτό το εμπόδιο θα υπερκεραστεί. Μέχρι το 2016 όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέος τελωνιακός κώδικας Προσβλέπουμε σε αυτό. Για την ώρα δημιουργούμε εθνικές ενιαίες θηρίδες. Θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία τον Ιούνιο του 2015. Απομένουν ακόμα εμπόδια για την εφαρμογή της οδηγίας όλα τα κράτη-μέλη, διότι οι εφορίες, οι φορολογικές αρχές έχουν ακόμα αφήσει τα εμπόδια να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τη διαβίβαση στοιχείων και την ασφάλεια όσον αφορά τα δεδομένα. Η ΕΜΣΑ πάντα πρόσεχε τα στοιχεία, έδινε σημασία στην προστασία των δεδομένων και όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται από την ΕΜΣΑ είναι ιδιοκτησία κυρίως των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να δίνουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς την άδεια των κρατών μελών ή της διευθύνουσας ε, ομάδας υψηλού επίπεδου, σε οποιονδήποτε βρίσκεται εκτός του πλαισίου αυτού, αυστηρότατος κανόνας που τηρούμε. Δεν δίνουμε πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος χωρίς την άδεια των κρατών μελών ή της διευθύνουσας ομάδας που ασχολείται με την ε, ασφάλεια των δεδομένων. Μετά Υπήρχε και άλλη ερώτηση για τις πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου και το κονδύλι που διατίθεται είναι περίπου 160,5 εκατομμύρια. Πριν είχαμε 154 εκατομμύρια, έχουμε μια αύξηση λοιπόν 6 εκατομμυρίων. Όμως βλέποντας τα νέα καθήκοντα που πρέπει να καλύψουμε, δηλαδή και τις πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ΕΜΣΑ. Τι κάναμε μέχρι τώρα. Δημιουργήσαμε ένα σχέδιο δράσης, πώς να αντιδρούμε σε περίπτωση ενδεχόμενου ατυχήματος που κανένας δεν θέλει να βλέπει, να δει, να συμβεί στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, με αυτά τα χρήματα είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περιέγραψα κάποια πράγματα στην παρουσίασή μου. Έχουμε συστήματα ε, ψεκασμού από αέρα και θα εξοπλίσουμε ένα-δύο σκάφη μας με δυνατότητα ψεκασμού ούτω ώστε να ψεκάζουμε ειδικέ ουσίες από τα σκάφη, την κοιλίδα και δημιουργούμε και αποθέματα για ψεκασμούς σε περιοχές όπου υπάρχουν ελλείψεις. Συνεργαζόμαστε πολύ με τη βιομηχανία του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ήταν πολύ θετική όσον αφορά τα όσα κάναμε και έχουμε άριστη ε, σχέση με, την, με τον τομέα και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών ΜΟΥΒ, Κριστίνα Μπέργκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα το τμήμα θαλασσίας ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, θαυμάσια συνεργασία που είχαμε και κατά την προηγούμενη θητεία με την Επιτροπή σας και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις που δεν απάντησε ο κύριος Μίλη γιατί δεν ε, αφορούν τις ε, απευθείας αρμοδιότητες της οργάνωσής του. Δεν χρειάζεται να πάτε στη Λισαβόνα για να μπορείτε να δείτε τα συστήματα πληροφορικής της ΕΜΖΑ. Έχουμε την 1η Δεκεμβρίου εδώ, σε ένα ξενοδοχείο, πίσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το βράδυ, μία παρουσίαση και μετά θα υπάρξει και μία δεξίωση. Εκεί μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας χωρίς να χρειαστεί να πάτε στην Λισαβόνα. Αν και καταλαβαίνω βεβαίω κύριε Μίλιο ότι με χαρά θα τους υποδεχόσασταν στη Λισαβόνα. Για τις ερωτήσεις. Για το θέμα του Φλαμίνια, το οποίο είχε απασχολήσει την Επιτροπή σας ε, την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο κύριος Μίλη. Τι έχουμε κάνει έκτοτε για να αποφευχθούν τέτοιες ε, περιπτώσεις. οι ανεξάρτητες αρχές ε, όλων των εθνικών κρατών που πρέπει να χορηγήσουν ε, θέση ασφαλούς λιμένα, που είναι θέμα μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, όλες αυτές συνεργάζονται και κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου με όλες αυτές τις οργανώσεις. Έρχονται εδώ λοιπόν και εξετάζουμε μια υποθετική περίπτωση, ένα πλοίο ζητάει βοήθεια και όλες οι αρχές που είναι παρούσες στο ίδιο σημείο, η πρώτη τέτοια άσκηση έγινε στο Ρότερνταμ, όλες πρέπει να δουν πώς θα, αποφύσουν, θα αποφασίσουν, πώς θα προχωρήσουν. Το πρόβλημα, ξέρετε, ήταν ότι το ατύχημα στο Φλαμίνια έγινε σε διεθνή ύδατα, οπότε ήταν ασαφές ποιος θα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία. Με βάση όμως τις ασκήσεις που κάνουμε, και τις λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούμε μαζί με αυτές τις αρχές εστιάζουμε κυρίως στην πρόληψη τέτοιων περιπτώσεων στο μέλλον. Είναι σχεδόν έτοιμες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και θέλουμε να τις ε, προωθήσουμε και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό γιατί αυτά τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε. Ίσως να ακούσατε να έχετε ακούσει και για την περίπτωση του Μέιζη όπου υπήρξε διαφωνία μεταξύ Νότιας Κορείας και Ιαπωνίας. Είναι λοιπόν παγκόσμιο θέμα. Έχει γίνει θαυμάσια εργασία λοιπόν στην Ευρώπη και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Επίσης, για το θέμα που μας ανησυχεί όλους. Θέλουμε Ευρωπαίους ναυτικούς Πρέπει να κάνουμε όμως μια διάκριση, διάκριση μεταξύ των βραχυπροθέσμων ενασχολήσεων με την ε, ναυτιλία όπου πηγαίνουν κάποιοι σε κάποια εκπαίδευση ή για μικρά χρονικά διαστήματα σε πλοία και μετά επανέρχονται. Εδώ έχουμε και περισσότερες γυναίκες ή ε, σε αντιπαράθεση με τους ναυτικούς ας πούμε ανοιχτής θαλάσσης που πολλές εβδομάδες λείπουν από τα σπίτια τους. Χάρη στην νομοθεσία που πέρασε κατά την προηγούμενη θητεία, δημιουργούμε μια βάση ενημέρωσης μαζί με την ΕΜΖΑ για να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τους ναυτικούς. Γιατί προς το παρόν αυτό είναι κύριο θέμα. Δεν ξέρουμε καν πόσοι Ευρωπαίοι είναι ναυτικοί σε πλοία με σημαίε των ευρωπαϊκών χωρών και σημαίε άλλων χωρών. Έχουμε κάποιε εκτιμήσει αλλά όχι ακριβή στοιχεία. Αυτό θα μα επιτρέψει μαζί με την τεχνολογία να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για να προσελκύσουμε περισσότερους νέους. Είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους νέους ναυτικούς, Ευρωπαίους. Για την έμπολα που έθιξε η κυρία Μάισναρ. Πρέπει να πω ότι χάρη στην υποβολή εκθέσεων από την ΕΜΖΑ και την ειδική μονάδα για το θέμα αυτό, την Task Force, πρέπει να πούμε ότι σε σχέση Εάν συγκρίνουμε με τις αεροπορικές ε, μεταφορές, είναι χαμηλού κινδύνου οι θαλάσσιες μεταφορές. Δεν έχουμε επιβάτες από τη Δυτική Αφρική, μόνο πληρώματα. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές από το από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όταν λοιπόν πλοία προσεγγίζουν τη Δυτική Αφρική δεν δίδεται άδεια αποβίβασης στο πλήρωμα για να μην υπάρξει κίνδυνος μόλυνσης. Και υπάρχουν και οδηγίες για τα πληρώματα που επιστρέφουν από αυτή την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο κλάδος να τηρεί τις προδιαγραφές για να μην υπάρξει οικονομική κατάρρευση στις χώρες έμπολα της Δυτικής Αφρικής γιατί δεν έχουν πλέον, αν δεν υπάρχουν θαλάσσιες μεταφορές για λόγους πρόληψης για παράδειγμα που μπορεί να φτάσει σε κάποια ε, ιστερική προσέγγιση θα έλεγα, μπορεί να υπάρξει λοιπόν αδυναμία των χωρών αυτών να εξάγουν. Θέλουμε λοιπόν σε επαφή με τον κλάδο να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση εάν κάποιοι, κάποιες εταιρείες, κάποιοι εφοπλιστές δεν θέλουν να προσεγγίζουν πλέον τα πλοία τους στις χώρες αυτές για να διατηρηθεί κάποια δυνατότητα οικονομικής σχέσης των χωρών αυτών με τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα για την ε, θαλάσσια χωρική, για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό, υπάρχει αυτή η οδηγία, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, να δούμε αν θα βοηθήσει. Σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους, να λάβουν στοιχεία για τις ε, διαδρομές των πλοίων ε, που υπάρχει συμφόρηση, συμφόρηση αλλά δεν έχει θεσμικό ρόλο της ΕΜΣΑ για, την, ε, για το χωρικό σχεδιασμό. Ελπίζω να κάλυψα όλα τα εναπομένοντα θέματα. Ευχαριστώ κυρία Μπέρκ, ευχαριστώ κυρία Μιλή. Οπότε κλείνει και το θέμα αυτό. Οπότε κλείνει η δημόσια συνεδρίασή μας. Α, η κυρία Μάισνερ. Ναι, πολύ σύντομα. Μιλήσατε για κατευθυντήριες γραμμές μετά το ατύχημα Έρικα πότε ακριβώς θα είναι έτοιμες, πότε θα μας αποσταλούν. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη φάση είναι σε φάση ολοκλήρωσης από τις εθνικές αρχές. Μετά θα κάνουμε διαβούλευση με τον κλάδο γιατί διάφορα τμήματα, για παράδειγμα, οι διασώστες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα λιμάνια, όλοι αυτοί πρέπει να δώσουν τη γνώμη τους Σωστό λοιπόν να δώσουμε και σε όλους αυτούς δυνατότητα να αντιδράσουν και όταν θα έχουμε την άποψή τους, αρχές της επόμενης χρονιάς, ελπίζουμε να καταλήξουμε. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Οπότε λίγη η εξέταση του θέματος αυτού. Τώρα θα έχουμε ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Αυτό όμως γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να παρακαλέσω τους επισκέπτες να αποχωρήσουν. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα η συμμετοχή σας. Σας εύχομαι ευχάριστη συνέχιση της παραμονής σας στις Βρυξέλλες.